We'll start the meeting and... Άρχεται η συνεδρίαση και μπορεί να τελειώσουμε και νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει, ελπίζω τουλάχιστον. Ας αρχίσουμε λοιπόν όμως με την οδηγία του Συμβουλίου και την εφαρμογή της ε, ε, Εφαρμογή τη οδηγία του Συμβουλίου 2078 τη 27 η Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, που συνήθως καλείται οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση. Έχουμε και προσκεκλημένου και θα αρχίσω δίνοντας το λόγο στην συγγνώμη, στην ε, υπηρεσία έρευνας και στο Χωσέ Λουίς Λούβας Κουιντάνα που θα μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα αυτό που έχουμε όμως συζητήσει και παλαιότερα στην Επιτροπή μας και ζητήσαμε να μάθουμε περισσότερα. Έχετε παρακαλώ το λόγο κύριε Κιντάνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία σύντομη ε, ενημέρωση προκειμένου να βάλουμε τα πράγματα στο πλαίσιο τους. Η Γενική Διεύθυνση ε, Υπηρεσιών Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βοηθά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου κάθε φορά που εξετάζουν ε, εκθέσεις εφαρμογής όπως και τώρα. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είχαμε προβλέψει μια, μια ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής που καλύπτει και τους τέσσερις λόγους ε, διάκρισης, διακρίσεων που προβλέπονται στην οδηγία, δηλαδή για λόγους θρησκείας, υπεπιθύσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσου προσανατολισμού. Το έγγραφο λοιπόν αυτό το οποίο σας δόθηκε εκπονήθηκε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την υπηρεσία αυτή έρευνας και έχουμε και ένα ακόμα έγγραφο, μια εξωτερική μελέτη αυτή τη φορά που εκπονήθηκε από την κυρία Χόλγουαρτ και η οποία έρευνα επικεντρώνεται στο πιο συγκεκριμένο ζήτημα των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεπιθήσεων, που είναι ένας από τους λόγους διακρίσεων που ανέφερα πριν από λίγο. Προτού όμως γίνει η που ειναι ενας απο τους λογους διακρισεων που ανεφερα από την κυρία Χόουαρτ, προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, ένα εισαγωγικό βίντεο το οποίο θα ήθελα να προβάλλουμε και συνέχεια θα μιλήσει η κυρία Χόουαρτ. Νομίζω ότι μπορούμε πάντως να δούμε τώρα το βίντεο πρώτα. Evaluation of its implementation. The European Union is founded on values such as respect for human dignity, freedom and democracy, and it shall combat social exclusion and discrimination. Employment is the most important condition for social inclusion. In 2000, the Employment Equality Directive was adopted in addition to the Racial Equality Directive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 Um, Καλό απόγευμα. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ε, οδηγία αυτή σε σχέση με τη θρησκεία και την πίστη. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε αυτόν τον λόγο διακρίσεων από άλλους. Υπάρχουν ε, κάποια θέματα που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με τη θρησκεία και την πίστη, αλλά και ε, άλλη πτυχή που έχει που έχει να κάνει με όλες τις διακρίσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω από δύο βασικά σημεία. Καταρχάς το ΔΕΚ πάντα υποστήριζε ότι εξαιρέσεις στην ίση μεταχείριση πρέπει να ερμηνεύονται πολύ στενά. Δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το απολύτως απαραίτητο οι εξαιρέσεις και θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά από το δικαστήριο. Η δεύτερη μου παρατήρηση έχει ιδιαίτερα να κάνει με τη θρησκεία και τις πεπιθήσεις. Ε, αυτός ο λόγος ε, διακρίσεων διαφέρει κάπως από τους άλλους λόγους, ε, διότι η ελευθερία στην θρησκεία και τις πεπιθήσεις προστατεύεται από τον ε, Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ε, και αυτό είναι σημαντικό διότι υπάρχει νομολογία υπό τη σύμβαση αυτή. Όχι όμως νομολογία του ΔΕΚ ακόμα. Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να μας βοηθήσει να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι η θρησκεία και οι πεπιθήσεις. Κάποιοι ε, υποστηρίζουν και καλύπτονται όντως ε, επειδή ε, γίνονται διακρίσεις εις βάρος τους επειδή δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη θρησκεία ή πίστη. Δύο θέματα εντοπίζονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014. Καταρχάς οι έμεσες διακρίσεις που έχουν να κάνουν με όλους τους λόγους ε, διακρίσεων που ε, αναφέρει η οδηγία στην πράξη, φαίνεται να είναι δύσκολη η εφαρμογή της ε, έννοιας αυτής. Οι έμεσες διακρίσεις πραγματοποιούνται Όταν ένας εργοδότης εφαρμόζει έναν ε, κανόνα που πρέπει να ισχύει για όλους τους εργαζομένους, ε, αλλά που κάποιοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν ε, λόγω της θρησκείας ή των πεπιθήσεων τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εργοδότης μπορεί να λέει ότι δεν επιτρέπεται να φοράει κανείς τίποτα στο κεφάλι στην δουλειά. Δηλαδή να φοράνε στολή. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για Εβραίους που θέλουν να φοράνε κήπα, για τις ε, μουσουλμάνες γυναίκες που φοράνε μαντήλα ή ε, για τους Σίκ που φοράνε τουρμπάνι. Σίχ. Και θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι αυτό τους εμποδίζει να πιάσουν δουλειά στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Αυτό λοιπόν μπορεί να αποτελεί έμεση διάκριση. Από την άλλη όμως θα πρέπει να εξετάσει κανείς εάν αυτή η διάκριση δικαιολογείται αντικειμενικά. Σύμφωνα με την οδηγία λοιπόν ο κανόνας θα πρέπει να έχει ε, θεμητό στόχο και θα πρέπει και τα μέσα για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ε, να ε, είναι αναλογικά. Το ΔΕΚ ισχυρίζεται ότι θα πρέπει αυτό να γίνεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, θα πρέπει τα μέσα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Δεύτερον, να είναι αναλογικά και να είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ο στόχος. Το δικαστήριο πάντα θεωρούσε ότι το απαραίτητα σημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί κανείς να πετύχει τον ίδιο στόχο με μέτρα που προκαλούν λιγότερες διακρίσεις. Παράδειγμα, ε, εργοστάσιο σοκολάτας ε, να έχει κανόνα ότι δεν επιτρέπεται οι άντρες να έχουν γένεια. Αυτό ισχύει για όλους. Ε, όσοι όμως ε, έχουν γένεια για θρησκευτικούς λόγους ε, δεν μπορούν να σπορφωθούν με τον κανόνα αυτό και έτσι δεν μπορούν να πιάσουν δουλειά στο εργοστάσιο. Αυτό φαίνεται να είναι έμεση διάκριση. Ε, ε, ε, δικαιολογείται. Ο στόχος είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων. Είναι θεμητός στόχος. Είναι όμως αναλογικό μέτρο το να πει κανείς ότι δεν επιτρέπεται να έχει γένεια να είναι αναλογικό μέτρο. Μπορεί να απαιτεί κανείς από τους άντρες να καλύπτουν τα γένια τους ώστε να μην γίνεται η διάκριση εις βάρος τους. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ο κανόνας αυτός όντως έμεση διάκριση. Και αναφέρομαι στη θρησκεία και τις πεπιθήσεις, αλλά ένα από τα πράγματα που έχει προκαλέσει δυσκολίες ε, στο πλαίσιο της ε, οδηγίας ήταν οι εξαιρέσεις από γενικές απαιτήσει για την απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας. Το άρθρο 4 ε, θεσπίζει κάποιε απαιτήσει, ε, για παράδειγμα, θεσπίζει κάποιες απαιτήσει σε περίπτωση που για παράδειγμα το φύλλο, η ηλικία ή κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο ε, για να κάνει κανείς αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει όμως αυτό να συνδέεται ε, με την ίδια τη δουλειά. Δεν μπορεί να έχει κανείς μια απέτηση πιο γενική. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητάει κανείς από κάποιον, ε, ζητάει κανείς ηθοποιό να παίξει τον Έλσον Μαντέλα σε μια ταινία μπορεί όντω να θέλει ε, έναν ε, μαύρο ηθοποιό, διότι είναι απαραίτητο αυτό. Για τι ε, θρησκείε όμω η οδηγία επιτρέπει άλλη μια εξαίρεση. Κάποιοι λένε ότι η εξαίρεση στο 4-2 είναι παρόμοια φύση. Έχει να κάνει με γενικέ προποθέσει απασχόληση. Και πάλι όμως συνδέεται με την φύση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ε, δουλειάς. Και λέει ότι δεν θα πρέπει να ε, ε, αιτιολογείται η διάκριση για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος θρησκευτικών σε ένα σχολείο να είναι ε, να είναι μουσουλμάνος. Ε, δεν μπορεί όμως να το ζητάει κανείς αυτό από τον καθαριστή, διότι δεν είναι απαραίτητο αυτό για να κάνει τη δουλειά του. Ε, επίσης δεν μπορεί να απορρίψει κανείς κάποιον επειδή είναι ομοφιλόφιλος, διότι και αυτό είναι διάκριση για άλλους λόγους. Κάποιοι έχουν πει ότι το άρθρο 4.2 δεν είναι απαραίτητο, καλύπτεται ήδη από το άρθρο 4.1. Υπάρχει και ένα άλλο μέρος του 4.2 που επιτρέπει από θρησκευτικούς οργανισμούς να ζητάει να είναι πιστοί οι άνθρωποι στη φιλοσοφία του Ιδρύματος αυτού, εφόσον όμως λέει ε, καλύπτονται οι άλλες προϋποθέσεις της οδηγίας. Το άρθρο αυτό δεν είναι πολύ σαφές. Ποιος ε, οργανισμός θεωρείται θρησκευτικός και η πίστη προς τον οργανισμό ε, πόσο μακριά πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά ή στην ιδιωτική ζωή του καθενός. Και επίσης ε, το να είναι κανείς ε, άθεος ε, ή να θεωρεί κανείς ότι το κράτος πρέπει να είναι κοσμικό είναι και αυτό μια φιλοσοφία στην οποία μπορεί να είναι κανείς πιστός. Όταν αξιολογούνται οι απαιτήσει που μπορίζει ένας ε, εργοδότης, ε, θα πρέπει να μπορεί κανείς ε, να τα εξετάσει αυτά και σε σχέση με την ισότητα, την αξιοπρέπεια και τις ανάγκες του καθενός. Θα πρέπει δηλαδή να εξετάσει κανείς τη γενική ισορροπία αλλά και με τις έμεσες διακρίσεις και με τις γενικές απαιτήσεις προς τους εργαζομένους. Αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ε, εξαιρέσεις ε, της οδηγίας και σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ε, έχουν εφαρμόσει όλα τα κράτη-μέλη τις εξαιρέσεις στο 4-2. Η Φιλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία δεν το έχουν εφαρμόσει. Σε άλλες χώρες όμως μπορεί να ερμηνευτεί το άρθρο 4.1 ώστε να καλύπτει τα θέματα του 4.2. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται κάποια επεξήγηση του ΔΕΚ. Το επόμενο ερώτημα όμως είναι εάν θα έχει την ευκαιρία το ΔΕΚ να ερμηνεύσει τα θέματα αυτά. Αυτό ήθελα να πω σχετικά με τη θρησκεία και τις πεπιθήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες αυτές παρατηρήσεις. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια Ρενάτε Βέμπερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την καθηγήτρια Χάουαρτ για τη μελέτη της. που εξέτασε την ε, εφαρμογή της οδηγίας ε, όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ε, ή υπεπιθύσεων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ε, Υπηρεσία Ερευνών μας ε, για τη δική της μελέτη, διότι ήταν πολύ χρήσιμες και οι δύο αυτές έρευνες ε, κατά την σύνταξη της έκθεσης που συζητάμε σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι, είμαι, ότι χαίρομαι πολύ που είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό, διότι το επάγγελμά μου σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάντα ασχολούμουν με το θέμα αυτό. Χαίρομαι λοιπόν που εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω τη δυνατότητα να εξετάσω το θέμα αυτό από διαφορετική οπτική. Το θέμα δηλαδή της απασχόλησης. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2015, φαίνεται περισσότεροι ε, Ευρωπαίοι να είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα θέματα διακρίσεων ομάδων και να είναι και καλύτερα ε, ενημερωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο σχετικό ευρωβαρόμετρο του 2012. Αυτό πιστεύω ότι αποτελεί πρόοδο σε κάποια κράτη-μέλη είναι καλύτερα ενημερωμένος ο κόσμος και επειδή τα ίδια τα κράτη-μέλη προχώρησαν πέρα από τις απαιτήσει της οδηγίας για την απασχόληση και δεν περιορίζουν τις διακρίσεις ε, στους τομείς ε, ε, της απασχόλησης ε, και της επαγγελματικής κατάρτισης, ε, αλλά καλύπτουν και τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία για τη Φιλετική Ισότητα. Ελπίζω ότι και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη στο μέλλον θα ακολουθήσουν την ίδια γραμμή. Ελπίζω ότι κάποια μέρα και η οριζόντια οδηγία ότι θα υπάρξει και οριζόντια οδηγία στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση. Δεν υπάρχουν ακόμα συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, όπως είχε οροματιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν προτάθηκε η οδηγία αυτή. Το σχέδιο έκθεσης, όσο έχει αυτή τη στιγμή, αποτελεί έκθεση πρωτοβουλίας και γνωρίζετε πολύ καλά ότι για το λόγο αυτό θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εκθέσεις αυτές. Έτσι λοιπόν ήταν ε, περιορισμένο το μήκος ε, της έκθεσης αυτής και νιώθω ότι είναι λίγο άδικο. Μέχρι 7 σελίδε μπορούσα εγώ να γράψω, ενώ εδώ έχουμε 70 σελίδες για το ίδιο θέμα. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε ότι όλοι οι συνάδελφοι θα συμβάλλουν σημαντικά με τις τροπολογίε που θα υποβληθούν. Είμαι πεπισμένη ότι στο τέλος η έκθεση αυτή θα έχει πολύ περισσότερο ψαχνό, να το πω έτσι, και ότι θα είναι πολύ πιο πλήρης. δεδομένου ότι η οδηγία καλύπτει τέσσερις λόγους διακρίσεων. Στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική και όσον αφορά ε, την ε, μορφή όσον αφορά τους διάφορους αυτούς τομείς. Πρέπει να πω ότι είχα αρκετές συναντήσεις με εκπροσώπους διαφόρων οργανώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, εταιριών. Και κατάλαβα ότι ναι, είναι καλό να έχουμε αυτούς, αυτούς τους τέσσερις λόγους διακρίσεως στην οδηγία, αλλά οι διακρίσεις που γίνονται στην πραγματική ζωή είναι πολύ διαφορετικές. Για παράδειγμα, όσον αφορά ε, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή ε, τη θρησκεία ή τις πεπιθήσεις. Σε κάποια κράτη-μέλη μπορεί να έχουμε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων οι οποίες όμως φαίνεται να είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Η καθηγήτρια Χάουαρτ μίλησε για τις έμεσες διακρίσεις. Και ναι, το βλέπουμε. Αυτό γίνεται μέσω νομοθεσίας που με την πρώτη ματιά φαίνεται ουδέτερη, αλλά έχει άλλες συνέπειες. Μετά έχουμε τις διακρίσεις λόγω ηλικίας που είναι πολύ πιο πολύπλοκες και φαίνεται να ε, να εμπεριέχεται συστημικά στην ομοθεσία μας, ώστε να μην το αντιλαμβανόμαστε καν ως διάκριση. Μετά από συναντήσεις που είχαμε εκπροσώπους ε, της κοινωνίας των πολιτών, φαίνεται ότι στην πράξη οι διακρίσεις λόγω ηλικίας συχνά ξεκινούν ήδη από την ηλικία των 40. διότι εάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε από τη μία τους νέους τους νέους άνεργους και από την άλλη από τα 40 και μετά ε, θεωρείται κανείς ε, υπερήλικας, ε, τότε πραγματικά θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα του ανθρωπίνου δυναμικού μας στην διεθνή αγορά. Όλα αυτά τώρα πώς ε, μεταφράζονται στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι δεν ε, νιώθουν ότι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κατάρτιση για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ε, δεξιότητες ή για να βελτιώσουν τις δεξιότητες που ήδη έχουν είναι οι πρώτοι που θα θεωρηθούν εξεπερασμένοι όταν η αγορά εργασίας θα αναζητάει νέες δεξιότητες και ας μην ξεχνάμε ότι η ψηφιακή αγορά ήδη είναι πραγματικότητα και σύντομα μάλλον θα μας ε, μεταφέρει σε νέους ορίζοντες. Από την άλλη μεριά, η πρόσβαση σε πρόορη σύνταξη έχει οδηγήσει σε στερεότυπα και επηρεάζει μέχρι και το 1 τρίτο των ε, ε, θέσεων, απασχόλησης, των πλήρους απασχόλησης. Σε περιπτώσεις αναπηρίας, όταν είναι εμφανής η αναπηρία, μιλάμε για μια κατηγορία ανθρώπων ε, που συχνά δεν δεν φαίνονται στην κοινωνία, είναι κρυμμένοι και θα έπρεπε να επενδύουμε σε ε, κοινωνικές πολιτικές που να επιτρέπουν την ένταξη των ανθρώπων αυτών. Κάθε φορά που εξετάζουμε την εφαρμογή της οδηγίας αυτής από τα κράτη-μέλη, αντιμετωπίζουμε έλλειψη ποιοτικών δεδομένων καθώς και ε, αντιμετωπίζουμε και την έλλειψη της υποχρέωσης των κρατών μελών να συλλέγουν ε, τα δεδομένα αυτά, κάτι αντιπαραγωγικό στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Έτσι είναι πιο δύσκολο αντικειμενικά να αξιολογούμε τις ε, εξελίξεις όσον αφορά την πολιτική και τις πρακτικές. Θέλω να πω σε λεπτομέρειες ε, σχετικά με το τι πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει για να αποφεύγονται οι διακρίσεις στον χώρο εργασίας. Ε, πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε όλα τα δικαιώματα και ότι θα πρέπει να έχουμε κοινωνίες με ποικιλομορφία. Η εναρμόνιση όσον αφορά τι διαδικασίε των κρατών μελών την ε, νομική εκπροσώπηση, την ε, νομική αρρωγή. Ε, χρειάζονται ακόμα κυρώσεις. Οι μηχανισμοί προσφυγής σε δικαστικές και μη δικαστικές αρχές θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε τα θύματα να έχουν πρόσβαση σε πλήρη αποζημίωση. Θα πρέπει να βοηθήσουν βοηθούνται οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οικονομικά μέσω διαφόρων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην προστασία των θυμάτων των διακρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την ενδυνάμωση των ανθρώπων με την ε, εκπαίδευση ε, μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων ώστε να ε, αναγνωρίζεται και να καταπολεμείται η ε, διάκριση εργαζομένων. Θα κλείσω εδώ και θα ήθελα πολύ να ακούσω τι έχουν να πούνε οι συνάδελφοι για τα θέματα αυτά. Ε, περιμένω να λάβω και τη συμβολή τους για την εκθεσία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους εσκιώδεις εισηγητές. Την κυρία Λόσκα Ράγεβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για την έκθεση αυτή την οποία έχει συντάξει. Πραγματικά το κείμενο αυτό βλέπουμε ότι άλλαξε πολύ από την τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε και βλέπουμε τώρα ότι πολλές από τις απόψεις που είχαμε εκφράσει στο παρελθόν έχουν ενσωματωθεί τώρα στην έκθεση. ευχαριστήσω λοιπόν για αυτό την κυρία Βέμπερ. Όχι τόσο η έκθεση, αλλά περισσότερο η οδηγία στην οποία αναφέρεται η έκθεση γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ιδίω όσον αφορά τη διάσταση των διακρίσεων λόγω θρησκείας υπεπιθύσεων. Ξέρετε ότι η Ευρώπη γίνεται όλο και πιο διαφορετική εμπεριέχει όλο και περισσότερους διαφορετικούς ανθρώπους, έχουμε όλο και περισσότερους μετανάστες και θα έχουμε και τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερους μετανάστες. Συνεπώς η οδηγία αυτή αλλά και άλλες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν σχέση με το ζήτημα αυτό, καλούνται αυτή τη στιγμή να επιλύσουν προβλήματα ή ακόμα και την ένταση που δημιουργείται σε πολλές χώρες και η οποία θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θεωρώ ότι οποιασδήποτε παρατηρήσεις ή τροποποιήσεις για την έκθεση αυτή που έχουν να κάνουν με τη θρησκεία, την πεποίθηση, την ανεξιθρησκεία κτλ. θα πρέπει να τονιστούν ακόμα περισσότερο, ακριβώς επειδή είναι ζητήματα όλο και πιο σημαντικά στο εφιστάμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακριβώς για τους ίδιους λόγους νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο το ζήτημα της διαφορετικής εκπαίδευσης που μπορεί να προσφερθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι τυπική είτε είναι άτυπη. Γιατί αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια νέα τάση που χαρακτηρίζεται από νεοφασιστικές τάσεις, από ξενοφοβία και συνειδητοποιούμε τελικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιεί το κόσμο και να γνωρίζει ποιε είναι οι βασικέ αρχέ και οι βασικοί κανόνε που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω τώρα κάποιε πιο λεπτομερεί παρατηρήσει. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, θα περάσω τώρα σε κάποιες πιο λεπτομερείς παρατηρήσεις. Το κεφάλαιο που έχει να κάνει με την αναπηρία. Καταρχάς, Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να επανέλθουμε στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να έχουμε και έναν ορισμό για το τι εστί άτομο με αναπηρία. Η Σύμβαση λέει ξεκάθαρα ότι η αναπηρία προκύπτει πολλές φορές ως αποτέλεσμα επαφής με το περιβάλλον, και το περιβάλλον αυτό μπορεί να αυξήσει, να μειώσει το βαθμό αναπηρίας ενός ανθρώπου. Και δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα μόνο στο επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά στο γενικότερο περιβάλλον. Και γίνονται εδώ πέρα κάποιες αναφορές σε αρχές οι οποίες υφίστανται πολλές φορές σε εθνική νομοθεσία. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε γενικό περιβάλλον να μπορεί να προκαλεί ή να δημιουργεί διακρίσεις και όχι μόνο το εργασιακό περιβάλλον. Έπειτα το κεφάλαιο που έχει να κάνει με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και συγκεκριμένα παράγραφος 16. Στην ε, παράγραφο αυτή γίνεται μία μία στο ότι ε, η ηλικία είναι ο πρώτο λόγο εισαγωγή διακρίσεων στον τομέα τη απασχόληση. Δεν είμαι πεπισμένη ότι όντω ισχύει κάτι τέτοιο. Αν πάρουμε αυτού του περίφημου τέσσερι λόγου διακρίσεων, Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι όντω η ηλικία είναι ο πιο σημαντικό παράγοντα στην Πολωνία, αλλά πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει και σε άλλε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, 90% ατόμων τα οποία είναι άνεργα, αλλά είναι άτομα με αναπηρίε. Δεν είναι απλώ άτομα τα οποία έχουν μια κάποια ηλικία. Έπειτα, όσον αφορά την αγορά εργασία πάλι, η ψηφιοποίηση, το νέο ψηφιακό περιβάλλον. Εδώ πέρα τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για τα άτομα με αναπηρίε, αλλά πρέπει να φερόμαστε εδώ πέρα στις γενικότερες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν όλο και πιο αποτελεσματικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένε αναφορέ στα προγράμματα κατάρτιση από τα οποία θα πρέπει να περάσουν οι άνθρωποι αυτοί, να μην αφαιρόμαστε στο ψηφιακό περιβάλλον ω απειλή, αλλά ω μια νέα ευκαιρία. Να μην χρησιμοποιούμε δηλαδή την ψηφιοποίηση, το ψηφιακό περιβάλλον ω πρόσχημα για να αποκλείουμε κάποιου ανθρώπου από την αγορά εργασία. Το πρόβλημα προφανώ δεν είναι το ψηφιακό περιβάλλον. Αυτό είναι θετικό και μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένοι εργοδότε χρησιμοποιούν το ψηφιακό περιβάλλον ω πρόσχημα για να αποκλείσουν κάποιου ανθρώπου από την απασχόληση, από το εργασιακό περιβάλλον. Όσον αφορά τώρα την παράγραφο 19. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στην επανεκπαίδευση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Και πάλι στο γενικότερο περιβάλλον των ψηφιακών δεξιοτήτων. Πάλι από αυτού θα ήθελα να πω ότι το σημαντικό δεν είναι εδώ πέρα οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι να επανεκπαιδευτούν, αλλά να διατηρήσουν και να βαθμίσουν κάποιε δεξιότητε του προκειμένου να καταφέρουν να διατηρήσουν τη θέση απασχολήσή του. Ακριβώ επειδή το ίδιο το εργασιακό περιβάλλον αλλάζει. Δεν λέμε ή δεν θα πρέπει να λέμε εδώ πέρα ότι απαιτείται κανεί να αλλάξει δουλειά εξαιτία του ψηφιακού περιβάλλοντο. Τώρα, το κεφάλαιο αυτό που έχει να κάνει με τον γενετήσιο προσανατολισμό πρέπει επίση να μα απασχολήσει. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να γίνονται αναφορέ και σε άλλε εκθέσει που έχουμε υποβάλει. Ακόμη και σε εκθέσει που έχουν υποβάλει διάφοροι εθνικοί φορεί ΛΟΑΔΜΑ. Στο σημείο 24 καλούμε τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν σαφείς ορισμούς για τον όρο μέλη της οικογένειας των οικογενειών ΛΟΑΔΜΑ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω σε τι αναφερόμαστε εδώ πέρα. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε λίγο το σημείο αυτό, προκειμένου να καταστεί λίγο πιο ξεκάθαρο. Και θα μπορέσουμε συνέχεια εμεί να πούμε στην εισηγήτρια να συμφωνούμε ή όχι με την παρατήρηση αυτή. Έπειτα, στο σημείο 28, στο κεφάλαιο οριζόντιες πτυχές και συστάσεις, γίνονται σαφώ πολύ θετικέ συστάσει στο έγγραφο αυτό. Λέτε όμω εδώ πέρα ότι τα θύματα θα πρέπει να χαίρουν φορολογικών απαλλαγών. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπερβάλλουμε λίγο. Πρέπει να αποσύρεται, πιστεύω, το σημείο αυτό και θα υποβάλω σχετικά και μια τροπολογία. Στη συνέχεια, δικαιολόγηση, αιτιολόγηση, άλλο σημείο στο κείμενο. Λέτε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ελάχιστες καταγγελίες κατά των διακρίσεων, γιατί πολλές φορές οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και γι' αυτό το λόγο δεν υποβάλλουν κάποιες καταγγελίες. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας ακόμα λόγος. Πολλές φορές τα άτομα τα οποία θεωρούν ότι είναι θύμα διακρίσεων θα υπέφεραν καταγγελία αν ε, πίστευαν ότι αυτό θα οδηγούσε κάπου, ότι θα οδηγούσε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το πρόβλημα τελικά έχει να κάνει με την ίδια την νομοθεσία, που ενδεχομένως δεν παροτρύνει τα άτομα να υποβάλουν καταγγελίε ακριβώς επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν την εργασία τους και γι' αυτό θα θέλουν να υποβάλουν μια τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Μπλενκεβιτσούτε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητριά μας, την κυρία Ρενάτε Βέβερ, διότι πραγματικά είναι πολύ καλή η έκθεσή της, πολύ καλά συνταγμένη και αν εργαστούμε ως ομάδα σε εργαστή συνεργασία θα την βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Ακούσαμε την αξιότιμη κυρία Χάουαρτ να μας κάνει την παρουσίαση της μελέτης που αναθέσαμε για τις διακρίσεις με βάση τη θρησκεία ή τις πεπιθήσεις. Θα ήθελα παρακαλώ να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια θέματα που αξίζουν τον κόπο να αναφέρονται στην έκθεση. Πρώτα απ' όλα η ηλικία. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρώπη γυράσκει. Ο κόσμος ζει περισσότερο και αναπόφευκτα θα δουλεύει και περισσότερο. Και ε, μετατίθεται προς τα πάνω ηλικία συνταξιοδότηση. Και αν δούμε τι γίνεται στα διάφορα κράτη-μέλη, θα διαπιστώσουμε πολύ εύκολα ότι οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν πάντα την ευκαιρία να παραμένουν στην αγορά εργασίας ή να εισέρχονται ξανά στην αγορά εργασίας μετά από κάποια διακοπή. Αυτό συνιστά διάκριση και ο κόσμος το νιώθει αρκετά και συχνά. Όταν για κάποιο λόγο κάποιος ακούει ότι καιρός είναι να πηγαίνει, να αποσύρεται για να ανοίξει θέση για κάποιο νεότερο. Το όπως τους νέους. Η οδηγία όμως κάτι τέτοιο το απαγορεύει. Εγώ δεν θέλω κανένα κοινωνικό αυτοματισμό ή να έρχονται γενιές αντιμέτωπες η μια στην άλλη. Η κάθε γενιά θα πρέπει να βρει τη θέση που της αναλογεί στην αγορά εργασίας και ο καθένας να έχει τις ευκαιρίες του στην αγορά εργασίας και να μην υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Ένα άλλο στοιχείο είναι η αναπηρία. Το πρωί συζητήσαμε πάρα πολύ τα θέματα αυτά, κυρίως τη σύμβασης ε, του ΟΗΕ για τους αναπήρους και πώς αυτή εφαρμόζεται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα πληθυσμού που υφίσταται διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Πρώτα απ' όλα, για λόγους πρακτικούς, οι χώροι δουλειάς δεν είναι συχνά προσαρμοσμένοι στις ανάγκες αυτών των ατόμων με αναπηρία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κατάφερε να ε, περάσει υποχρεωτική δεσμευτική νομοθεσία σχετικά. Βέβαια αυτό χρειάζεται επενδύσεις στους χώρους δουλειά για να προσαρμοστούν και να συντρέχουν εκείνοι οι ε, λόγικοι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία να εργάζονται. Εξάλλου, τα άτομα με αναπηρία δεν έχουν αρκετά κίνητρα για να μπουν στην αγορά εργασίας. Η επαγγελματική κατάρτιση συχνά είναι ανύπαρκτη για ανθρώπους με αναπηρία. Και εδώ χρειάζεται ε, συνεργασία με τους εργοδότες και γενικότερα με όλους τους ενεχομένους φορείς και τους ίδιους αναπήρους και τις οργανώσεις τους για να δούμε πώς ε, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην αγορά εργασίας. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να το κάνουμε και στην έκθεση να ε, προβεί σε μια αναθεώρηση ενδιάμεση της στρατηγικής για τους αναπήρους 2010-2020. Κάτι άλλο που ανέφερε η συγγήτρια και το λέει και η έκθεση είναι η συλλογή στοιχείων και δεδομένων. Γιατί δεν το επιτρέπει αυτό η οδηγία. Δύσκολα να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να έχει δεδομένα και στοιχεία στη διάθεσή του. Το ξέρω ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών αυτή, αλλά θα πρέπει να καλέσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη ζητήσουμε να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η συλλογή στοιχείων στα κρατη Στην έκθεση θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί το θέμα της παρενόχλησης ε, στην εργασία και στον χώρο δουλειάς. Παρενόχληση για διάφορους λόγους. Ε, για λόγους σεξουαλικής ε, προτίμησης, ε, ηλικίας, φιλής, φίλου κλπ. Και χρειάζεται ιδιαίτερη πρόνοια και μέρημνα για την υποστήριξη που παρέχεται στα θύματα της παρενόχλησης. Ο κόσμος συχνά φοβάται όταν υφίσατε διακρίσεις για διάφορου λόγους, θρησκεία, ηλικία, γενετήσιο προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο φύλλο. Ο κόσμος φοβάται να υποβάλει κάποια καταγγελία, μην τυχόν και χάσει τη δουλειά του. Αυτό θέλει προσοχή και αύξηση της συνειδητοποίησης. Θα πρέπει να κοιτάμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Γιατί τα κράτη-μέλη μας έχουν διαφορετικές εμπειρίες από χώρα σε χώρα. Είμαστε 28 χώρες, ο καθένας έχει τις παραδόσεις και τις ε, συνήθειες. Δεν θα πρέπει κανείς να φοβάται να μιλάει για τις διακρίσεις που υφίσταται, εφόσον έχουμε αυτή την οδηγία. Ούτε να φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά του. Βέβαια χρειάζεται πάντα συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μεταξύ μας εμείς οι συγγητέ και σκιώδεις συγγητές για να βγει ένα καλό έγγραφο τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Χέλκα Στέβενς είναι σκιώδη συγγητρία και εκείνη. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαιρετίζω την έκθεση της κυρίας Βέμπερ. Εκτιμώ ιδιαίτερα τα όσα λέει και είναι πολύ θετική και η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε σήμερα το πρωί όσον αφορά τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι ε, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την αναφορά που γίνεται στη σύμβαση αυτή, στην ίδια την έκθεση και στις συστάσεις της σύμβασης αυτής. Θα ήθελα να αφαιρθώ στο κεφάλαιο αυτό που έχει να κάνει με την απειρία. Είναι ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και περισσότερα στοιχεία για τις μη προσαρμογές που δεν λαμβάνουν χώρα στο χώρο εργασίας για τα άτομα αναπηρία. Πιστεύω ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία ιεράρχηση όσον αφορά τις διάφορες μορφές διακρίσεων και ανησυχώ ιδιαίτερα για την πολλαπλή διάκριση που δέχονται ορισμένοι άνθρωποι. Νομίζω ότι εδώ πέρα χρειαζόμαστε περισσότερη νομική βεβαιότητα και νομική ασφάλεια. Και πολλές φορές υπάρχουν εδώ πέρα διαφορετικές προϋποθέσεις, διαφορετικοί κανόνες, κατακαιρματισμένο νομικό πλαίσιο στα κράτη-μέλη, πράγμα το οποίο δεν το αναφέρουμε στην έκθεση. Έχει αυξηθεί η σωρευμένη εμπειρία που έχουμε όσον αφορά την παρενόχληση και τη διάκριση. παρόλα αυτά όμω θα πρέπει να καταβάλλονται περισσότερα στοιχεία. Προκειμένου λοιπόν να εφαρμόζεται καλύτερα η οδηγία αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να αυξήσουμε το βαθμό ευαισθητοποίηση όσον αφορά την παρεχόμενη προστασία. Να έχουμε καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων προτού δημιουργήσουμε νέου κανόνε. Για παράδειγμα, να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τα εθνικά συστήματα καταβολή καταγγελιών και να έχουμε και την κατάλληλη λειτουργία των αρμοδίων φορέων στα κράτη-μέλη. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις των συναδέλφων και Χαίρομαι που βλέπω ότι οι φορείς καταπολέμησης των διακρίσεων έχουν λάβει μέρος και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος στην επεξεργασία της έκθεσης αυτής. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια καταπολέμηση διακρίσεων όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης, αλλά σε όλους τους κλάδους, όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Στίβενς. Το λόγο τώρα έχει η Ρίνα Ρόνια Κάρη, η οποία μου συναπούσα από ό,τι βλέπω. Άρα περνάω κατευθείαν στην Τατιάνα Στάνοκα, που είναι και αυτή σκιώδη εισηγήτρια. Έχετε το λόγο εξ ονόματο των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ρενάτε για την εξαιρετική της αυτή έκθεση. Και βέβαια να ευχαριστήσω και όλους όσοι συνέβαλαν στην έκθεση αυτή και ήδη βλέπουμε ότι η Ρενάτα έχει λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις που είχαμε υποβάλει στο παρελθόν, καθώς επίσης και τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι δύο προσκεκλημένοι μας που συνέταξαν την έρευνα που μας παρουσιάστηκε. Είναι πολύ καλαδομημένη η έκθεση αυτή. Έχουμε δύο εισαγωγικά σημεία όπως βλέπετε. Συμφωνώ 100% μαζί τους η έκκληση καταρχάς αυτή που γίνεται να βγούμε από το υφιστάμενο αδιέξοδο, το οποίο έχει δημιουργήσει προφανώς το Συμβούλιο, όσον αφορά μια οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, θα πρέπει συνεχώς να λέμε στο Συμβούλιο ότι μπορούν να το κάνουν αν θέλουν και ότι αυτή τη στιγμή δεν υπήρξε απαραίτητη πολιτική βούληση για να γίνει κάτι τέτοιο. Επίσης, αναφερθώ στο σημείο παριθμών 1 της έκθεσης που λέγεται ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμπεριλάβει συγκεκριμένες διατάξεις στην νομοθεσία τους. Παρ' όλα αυτά δεν καλύπτεται πλήρως το κείμενο της έκθεσης αυτής σε όλες τις εθνικές νομοθεσίες. Τώρα, όσον αφορά το σημείο 4. πιθανοί λόγοι διακρίσεων που καλύπτονται από την έκθεση. Μιλήσαμε αρκετά πιστεύω για τη θρησκεία και τις πεπιθήσεις. Έχουμε καλύψει επαρκώς το κεφάλαιο αυτό. Ακούσαμε και τις δύο μελέτες. Δεν έχω να πω επιπλέον πράγματα, απλώ το σημείο 4 της έκθεσης νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε λίγο τη διατύπωση. Ενδεχομένως να επαναδιατυπώσουμε το σημείο εκείνο που αναφέρεται στις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προφανώς χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες προς αυτό. Και να διαχωρίσουμε το σημείο αυτό από τις αποφάσεις που λαμβάνει το δικό μας το δικαστήριο, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Όσον αφορά τώρα το κεφάλαιο της αναπηρίας, η κυρία Στίβεν κάλυψε πλήρως το κεφάλαιο αυτό, αναφέρθηκε όμως αυτό και η Ρενάτε, το καλύψαμε πλήρως επίσης και με τη σημερινή μας πρωινή συνεδρίαση και στην έκθεση επίσης της κυρίας Στίβενς ε, έχουμε καλύψει το ζήτημα αυτό. Την αφερθήκαμε δηλαδή στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες. Όσον αφορά πάντως το κεφάλαιο αυτό στην έκθεση της κυρίας Βέμπερ, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δούμε πώς οι δικές μας συστάσεις, και από τις δύο εκθέσεις δηλαδή, θα μπορούσαν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να αποφύγουμε πιθανές αντιφάσεις. Ενδεχομένως θα ήταν θετικό να επαναλάβουμε εδώ πέρα και κάποιες από τις συστάσεις που έχουμε κάνει σε άλλες εκθέσεις. Όσον αφορά τώρα το κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ηλικία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες τροποποίησεις. Ξεχάσαμε εδώ πέρα να κάνουμε μία αναφορά στην απασχόληση. Ξέρω ότι έχουμε απασχόληση των νέων συγκεκριμένα, ανεργία των νέων. Ξέρω ότι έχουμε μία συγκεκριμένη έκθεση για το ζήτημα αυτό. Πάντως νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη μνήα στην ανεργία και ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων. Ω και ο Δεσηγήτρια είχα συνεργαστεί και για την έκθεση Κούκαν, όπου αναφερθήκαμε στον ενεργό γυράσκοντα πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρετε ότι είχαμε και το έτος 2012 αφιερωμένο στο ζήτημα αυτό. Γίνανε κάποιες πολύ θετικές συστάσεις, μία εκ των οποίων ήταν να θίξουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό σε ισότιμο επίπεδο με το πρόβλημα της ενεργείας των νέων. Θεωρώ ότι αναφερόμαστε πάρα πολύ συχνά στην ανική ενεργεία, πολύ θετικό αυτό, αλλά νομίζω ότι εξίσου θα πρέπει να αναφερόμαστε και στην ενεργία των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων. Άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, απέχουν 10 χρόνια από τη συνταξιοδότηση. Νομίζω ότι και αυτό το ζήτημα είναι εξίσου σημαντικό και θα πρέπει να το αναδείξουμε εξίσου με το πρόβλημα της δανεικής ανεργίας και προφανώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με απόλυτη σοβαρότητα και σχετική μνήμα θα πρέπει να γίνεται βέβαια και στην έκθεση αυτή. Ας περάσουμε τώρα στο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το γενετήσιο προσανατολισμό. Συμφωνώ απόλυτα ότι το σημείο 24 θα πρέπει να αποσαφινιστεί λίγο περισσότερο. Μέλη της οικογένειας των οικογενειών ΛΟΑΔΜΑ. Στη δική μου εκλογική περιφέρεια η οικογένεια εννοείται ως οικογένεια μεταξύ άνδρας και γυναίκας, άνδρα και γυναίκας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε πώς κράτη-μέλη με διαφορετική εθνική νομοθεσία μπορούν τελικά να καταλήξουν σε έναν σαφή ορισμό για τον όρο μέλη της οικογένειας των οικογενειών ΛΟΑΔΜΑ. Καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε διάκριση στην δική μας εθνική νομοθεσία, προτού βελτιώσουμε τις νομοθεσίες αυτές. Σχετικά λοιπόν εγώ θα υποβάλω μια τροπολογία, δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο περιέγραψε ισχύει μόνο για την Λετωνία. Ανάλογα φαινόμενα πιστεύω ότι έχουμε και σε άλλες χώρες όπως η Λιθουανία. Τώρα, όσον αφορά το κεφάλαιο οριζόντιες πτυχές και συστάσεις, θα ήθελα να αφαιρθώ εδώ πέρα στην ποιότητα των δεδομένων, στα ποιοτικά δεδομένα. Πολλοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι έχουμε καταρχάς μία απουσία δεδομένων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εσύ Ρενάτε λες εδώ πέρα ότι ε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμος να προωθήσει τη συλλογή δεδομένων, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό σύσταση στο διατακτικό, όχι μόνο στα εκτιμώντας όπως τώρα το αναφέρεις. Έχουμε όμως και τα δεδομένα από τη Eurostat, έτσι δεν είναι. Εγώ υπήρξα εισηγήτρια συντάξει μιας έκθεσης για τα ad hoc μοντέλα, τα ad μοντέλα συλλογής δεδομένων από τις στατιστικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη Eurostat. Και τότε οι περισσότερες πολιτικές ομάδες δεν είχαν δεχθεί την πρότασή μου να συμπεριληφθούν και τα δεδομένα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με την εμφάνιση διακρίσεων λόγω θρησκείας πεπιθήσεων, γενετήσου προσανατολισμού ή λόγω φιλής ή λόγω ε, φιλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ζητήματα που καλύπτονται από άλλες οδηγίες. Είχα πει τότε ότι θα έπρεπε να συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα και για αυτά τα ζητήματα. Και μάλιστα είχα δει τότε πώς λειτουργούσαν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και είχα συνειδητοποιήσει ότι ε, ορισμένες μόνο τέτοιες στατιστικές υπηρεσίες συνέλεγαν τα δεδομένα αυτά κατά τρόπο εθελούσιο όμως, δεν υπήρχε υποχρεωτική δέσμευση. Κάποιες στατιστικές υπηρεσίες είχαν και κάποια ερωτηματολόγια για τα ζητήματα αυτά. Εγώ είχα πει τότε ότι θα έπρεπε να είχαμε κοινά τέτοια ερωτηματολόγια για όλες τις στατιστικές υπηρεσίες και να προβλέπεται μια πανευρωπαϊκή συλλογή τέτοιων δεδομένων. Ας μας, α, ας μας απασχολήσει αυτό τουλάχιστον στο μέλλον ώστε να καταφέρουμε να έχουμε τελικά δεδομένα για πιθανές μορφές διακρίσεων. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, madam. Ε, ευχαριστώ, κυρία μου. Θα δώσω το λόγο στη Λάουρα Τζέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη συνάδελφο Βέμπερ. Διότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η εισηγήτρια προσπάθησε πραγματικά να επικεντρωθεί στη μεγαλύτερη δυναμία της οδηγίας αυτής. Γινόταν λόγος για τις διακρίσεις, και αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά εδώ μιλάμε κυρίως για το ζήτημα της εφαρμογής οδηγίας στον τομέα της απασχόλησης. Η οδηγία πολλές φορές απλώς περιοριζόταν στο να καταγγείλει τους διάφορους τύπους διάκρισης, χωρίς όμως να προβλέπει μία ανάλυση των διακρίσεων αυτών στον τομέα της απασχόλησης. Νομίζω λοιπόν ότι με την έκθεση αυτή σημειώνεται ένα σαφές βήμα πρόοδου και μπορούμε πραγματικά να εστιαστούμε ουσιαστικά στο ζήτημα των διακρίσεων στον χώρο της απασχόλησης. Υπάρχουν βέβαια εδώ κάποια δύναμα ακόμα σημεία, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε κάποιες βελτιωτικές τροποποίησεις μέσω τροπολογιών. Για παράδειγμα, κάνετε δύο αναφορές τις οποίες πρέπει να αναλύσουμε λίγο περισσότερο πιστεύω. Όταν για παράδειγμα λέτε ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε προσαρμογές στο χώρο απασχόληση προκειμένου να μην γίνονται θύματα διακρίσεων τα άτομα με αναπηρίες. Προφανώ αυτό είναι πολύ σημαντικό αλλά νομίζω ότι θα πρέπει επ' αυτού να υπάρχει και η απαραίτητη νομική βεβαιότητα, νομική ασφάλεια. Ένα άλλο σημείο στο οποίο πιστεύω ότι πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο είναι η γενικότερη προσαρμογή του χώρου απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία. Είχα συμμετάσχει στο παρελθόν σε μία σχετική έκθεση και είχα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και σήμερα το πρωί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συζήτηση που έγινε όσον αφορά την ε, αναπηρία, τα άτομα αναπηρία και πιο συγκεκριμένα στο χώρο της απασχόλησης, όχι μόνο δηλαδή να δούμε πού εμφανίζεται η διάκριση και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά πέρα από αυτό να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε και εμείς, αν θέλετε, ένα όραμα, μια πιο συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Κάποιες επιμέρους ακόμα παρατηρήσεις θα μπορούσα να κάνω για άλλα σημεία, αλλά νομίζω ότι αξίζει να εμβαθύνουμε περισσότερο στα σημεία τα οποία έθιξα και για τα οποία θα υποβάλω και τροπολογίες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την κοινωνική προστασία των ανθρώπων ποια είναι η αποζημίωση που θα προβλέπουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης ή η προσβαση στις θέσεις απασχόλησης, ποιες είναι οι εθνικές διατάξεις όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης. Όλα αυτά είναι σημεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για τα οποία αυτή τη στιγμή η έκθεση είναι κάπως παρουσιάζει μια κάποια δυναμία και είναι σημεία τα οποία τελικά δεν διευθετεί ούτε η οδηγία, τα έχει παραβλέψει εντελώς. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτά τα σημεία και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές μορφές διακρίσεων. Συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφος πριν από λίγο όσον αφορά το ζήτημα της παρενόχλησης στον χώρο της απασχόλησης. Υπάρχουν πάρα πολλές και διαφορετικές μορφές διακρίσεων. Ας μην περιοριζόμαστε όμως στο να καταγγείλουμε μόνο τι διακρίσεις αυτές. Ας κάνουμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης τους. Ας δημιουργήσουμε ένα κάποιο ευρωπαϊκό όραμα για την αντιμετώπιση των διακρίσεων αυτών πολλές φορές δεν γίνονται καταγγελίες ακριβώς επειδή δεν γνωρίζουν τελικά οι ίδιοι οι φυγόμενοι πώς θα προστατευθούν τα δικαιώματά τους. Και σε σχέση και με μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε την Ιρανάτε να θίξω ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο ελπίζω ότι θα λάβει υπόψη τη συζητήτρια. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια επίγουσα κατάσταση αυτή της μετανάστευσης, του προσφυγικού ζητήματος. Προσπαθούμε όλο και περισσότερο να ενσωματώσουμε τους πρόσφυγες στην αγορά εργασίας. Πώς μπορούμε εκεί να αποφύγουμε τις διακρίσεις. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ενσωμάτωση των μεταναστών στο χώρο εργασίας θα γίνει χωρίς την εμφάνιση διακρίσεων κατά των προσφύγων. Χωρίς δηλαδή να προκύψει ακόμα μία παραπάνω ρήξη, αν θέλετε, ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους που προσπαθούν αυτή τη στιγμή να ενσωματωθούν ο ένας στον άλλον. Σε ευχαριστώ πάντο, πάρα, πάρα πολύ Ρενάτε πάντως για την έκθεσή σου αυτή, γιατί πραγματικά η οδηγία είχε πολλά κενά, πολλά σαφή σημεία και ξέρω ότι εσύ προσπάθησες μέσω της έκθεσής σου αυτής να καλύψεις όλα αυτά τα κενά. Ευχαριστώ πολύ. Μάρα Πισότ. Όχι, κύριε Μαρτέν, κύριε Μαρτέν, δεν έδωσα το λόγο σε εσά. Α, καλά. Μιλήστε. Λοιπόν, διάκριση στην απασχόληση σε σχέση με τη θρησκεία, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Άκουσα τις κυρίες Χάουαρτ ε, Βέμπερ και κάποιους από τους σκιώδεις ηγητές. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία εδώ και ένα πρόβλημα. Άλλος φοράει Κήπα, άλλος τουρμπάνι, άλλη μαντήλα, άλλος έχει μουσι. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Ότι θέλουν να τους ικανοποιήσουν όλους αυτούς. Και δυστυχώς αυτή η λύση είναι λάθος δρόμος, στραβός και λάθος και αδύνατο. Η λύση θα περάσει μόνο από αυτό που στα γαλλικά λέγεται λαϊσιτέ, το κοσμικό χαρακτήρα του κράτους δηλαδή. Οφείλει το κράτος να είναι κοσμικό και η μόνη κοινότητα που αναγνωρίζεται με αλφαγιώτα είναι ε, η εθνική, δηλαδή όλος ο λαός. Η θρησκεία θα πρέπει να ανήκει στην ιδιωτική σφαίρα και μόνο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβάλλεται ε, με τρόπο εμφανή και επιδεικτικό στους υπολείπους πολίτες. Όλοι γνωρίζουν ότι η ελευθερία όλων αρχίζει εκεί που σταματάει η ελευθερία των άλλων. Μόνο έτσι και μόνο έτσι θα μας απλούστευε πολύ τη ζωή μας. Ούτε κύπα, ούτε τουρμπάνι, ε, ούτε μαντίλα, ούτε τίποτα, ούτε ε, μουσι σε κανένα επάγγελμα. Το ίδιο ισχύει και για το γενετήσιο προσανατολισμό. Είναι προφανές ότι αυτό ε, είναι κάτι που ανήκει στην ιδιωτική ζωή του καθενός και δεν χρειάζεται να την επιδεικνύουμε δημοσίως. Προσωπικά δεν είδα δημόσια εκδήλωση σε άρματα ετεροφιλοφίλων που να ε, χορεύουν γυμνοί και να μιμούνται τη σεξουαλική πράξη. Όχι απλώς είναι αυτό η ιδιωτική ζωή, αλλά μάλιστα είναι ε, και θέμα που αφορά την κρεβατοκάμερα και μόνο. Κάποιος έλεγε για τη μητέρα των σπίτι, δεν θα φανταζόμουν ποτέ αυτή, αυτή η γυναίκα με τα άσπρα μαλλιά ε, θα ήξερε πώς γίνονται τα παιδιά. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ ιδιωτικά και σε ό,τι αφορά την ε, ηλικία, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν εργοδότες και είστε υποχρεωμένοι να το δεχτείτε, δεν ξέρω πώς θα το καταπολεμήσετε, ότι ένας εργοδότης πάντα, τουλάχιστον σε θέματα που έχουν σωματική δραστηριότητα και χρειάζονται δύναμη, ο πάντα θα προτιμά ένα νέο που θα είναι και πιο αποδοτικός και θα του κοστίζει λιγότερο από ένα μεγαλύτερο που θα έχει χαμηλότερες επιδόσεις και θα είναι και πιο ακριβώ. Δεν ξέρω πώς θα το παρακάμψετε αυτό το ζήτημα που είναι κάτι το προφανές και το αυτονόητο. Η κυρία Μπιζότο τελικά για το θέμα των αναπήρων μου ζήτησε να σας πω τα Να επιμείνω στο γεγονό ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί κάθε είδου διάκριση ε, που να εμποδίζει την πλήρη ένταξη των αναπήρων στην αγορά εργασία. Γιατί υπάρχουν εμπόδια και φυσικά, δηλαδή όχι νομικά εμπόδια, κανονικά εμπόδια, ε, άμεσα αλλά και έμεσα. Επιμένει επίση την έλλειψη συστημάτων κατάρτιση και ειδική σταδιοδρομίας μαζί ε, με την αγορά εργασία, μετά από συνεννόηση. Αυτά τα είπανε διάφοροι και τα έχουν ξαναπεί. Τελικά συμφωνούμε για να μπορούν οι ανάπηροι να αναπτύσσονται, να ε, ανθίζει προσωπικά τους με αυτονομία. Και τέλος, και εν κατακλείδη, όπως και εσείς φυσικά, εμείς θα υπερασπιστούμε τη γενική αυτή αρχή, ίση αμοιβή για ίση εργασία χωρίς καμία διάκριση κανενός είδους. Στο βαθμό που οι άνθρωποι ξέρουν να σέβονται την ελευθερία των άλλων και να αφήνουν την ιδιωτική σφαίρα στην απόλυτα ιδιωτική ζωή του καθενός. Ευχαριστώ. Thank you, Madam. Ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο η κυρία Λόπες Φοντανιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Βέμπερ για τη σπουδαία δουλειά που έχει κάνει. Επτά σελίδες μπορεί να είναι, αλλά πάρα πολύ συμπυκνωμένες και πάρα πολύ μεστές και λένε την κεντρική ιδέα. Όταν γίνεται λόγος για διάκριση, ε, διακρίσεις γίνονται στη δουλειά και το ξέρει ο πληθυσμός και η κοινωνία. Όπως είπε η όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ε, ξενόφοβες δηλώσεις, ομοφοβικές ε, που έχουν αυξηθεί με τις μεταναστευτικές και προσφυγικές κρίσεις. Και εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθούμε τις αρχές μας και να αυξήσουμε τις ε, δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για να σταματήσει η ε, ρίζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας μας. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ στα εξή δύο σημεία και δύο ομάδες που θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στο κείμενο. Πρώτον, το είπε και η κυρία Κοσλόφ Καραζέσκη, ε, μίλησε για την κοινότητα των Ρωμά. Είναι εθνική μειονότητα ε, που κινδυνεύει πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ διαδεδομένη. Στην Ισπανία έχουμε πολλούς και ο αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας είναι άνω του 78%. Το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό και τα μέτρα που χρειάζονται βράχει πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και υποστήριξη των ΜΚΟ. Και πολλές από τις ΜΚΟ είναι των ίδιων των Ρωμά που είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα το πρόβλημα, την πραγματικότητα και μπορούν φυσικά να βοηθήσουν καλύτερα τους δικούς τους ανθρώπους. Και επίσης γίνεται μεγάλος λόγος για τους ανθρώπους με αναπηρία. Εγώ μάλιστα θέλω να μιλήσω για τις γυναίκες της ανάπηρης, διότι αντιμετωπίζει διπλή διάκριση αυτή η κατηγορία πληθυσμού, για να μην πω και τριπλή όταν ανήκουν και σε εθνική ε, μειονότητα ή είναι μετανάστριες. Εκεί η απασχόλησή τους είναι κάτω του 50%. Χρειάζονται δηλαδή προσαρμογές στην αγορά εργασίας και αυτό είναι ένα μόνο βήμα, ένα πρώτο βήμα για να βελτιωθεί ε, η ένταξη και η ε, λεγόμενη απασχολησιμότητα των αναπήρων και να γεφυρωθεί το χάσμα του φύλου. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό. Να επιμείνουμε, επαναλαμβάνω, στην εκστρατεία ενημέρωση, πληροφόρηση, τα δικαιώματα των δύο αυτών ομάδων. Καλύτερη συλλογή δεδομένων και στοιχείων για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και να αναλύουμε καλύτερα πώς εφαρμόζεται η οδηγία και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Σούλτσε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια. Ακούσαμε πολλούς που μακρηγόρησαν. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τέσσερις παρατηρήσεις έχω. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση, διότι κατά τη γνώμη μου είναι πολύ ισορροπημένη και που θίγει πολλές σημαντικές πτυχές ε, πιο πολύ. Νομίζω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε την ψηφιοποίηση ώστε να αποτελεί ευκαιρία και για τους πιο ηλικιωμένους. Στο σημείο 18 μπορείτε να το βρείτε αυτό τουλάχιστον στην γερμανική μετάφραση. Βρίσκω πολύ αρνητική την διατύπωση. Ίσως θα πρέπει να φροντίσουμε η σχέση ανθρώπου με τα ρομπότ να αποτελεί ευκαιρία ώστε με την υποστήριξη των ρομπότ να μπορούν να παραμένουν περισσότερο στην αγορά εργασίας οι άνθρωποι. Το τρίτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο της οδηγίας. Είναι δύσκολη η συλλογή αυτή, συχνά πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα και είναι δύσκολο να βρεθεί ισορροπία ανάμεσα στην προσπάθεια που απαιτείται για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία και το αποτέλεσμα. Τέταρτη παρατήρηση στον αγώνα κατά των διακρίσεων. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η σύσταση που γίνεται εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Θα ήθελα να ακούσω εάν υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να θέλει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσής της, το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αναφέρεται σε ένα θέμα πολύ σημαντικό και για μας και για το οποίο έχουμε επενδύσει πολύ σημαντικές προσπάθειες. Ξέρετε ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των παραβιάσεων κατά της οδηγίας αυτής και προσπαθούμε και εμείς να προωθήσουμε προγράμματα ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα τα οποία θίξατε. Οποιαδήποτε λοιπόν υποστήριξη και από εσά είναι πρόσδεκτη. Καταγράφουμε προφανώς όλα τα ερωτήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά το ζήτημα των διακρίσεων λόγω θρησκείας υπεπιθύσεων. Προφανώς χρειαζόμαστε εδώ πέρα διευκρινήσεις και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως για τις εκκρεμείς υποθέσεις, και οι οποίες θα αποτελέσουν προφανώς, εφό όταν εκδικαστούν, ε, μέρος της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι ακόμα το οποίο προφανώς το γνωρίζει η δική σας η Επιτροπή, όσον αφορά την ε, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα των ε, καταπολέμησης των διακρίσεων κατά της αναπηρίας, έχουμε το, την πράξη αυτή της προσβασιμότητας, την οποία αναφέραμε και στην πρωινή συνεδρίαση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ενδεχομένως θέλει να συνοψίσει τη συζήτηση η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα τυχερή θεωρώ, γιατί ε, από κοινού εργαζόμαστε για την έκθεση αυτή με τους και οδησηγητές αλλά και με άλλους ε, συναδέλφους, με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσεγγίζουν τα πράγματα με το ίδιο πνεύμα και που ουσιαστικά ποθούν όλοι οι διακρίσεις να καταργηθούν, να μην θεωρούνται σε καμία περίπτωση αποδεκτές σε κανένα κράτος μέλος και πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι λοιπόν πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι στη θέση αυτή της εισηγήτριας και προσβλέπω σε περισσότερη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Μερικές μόνο σύντομες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω επί του παρόντος γιατί ξέρω ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε περαιτέρω την έκθεση αργότερα. Όσον αφορά τις συστάσεις, που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή και τις άλλες συστάσεις που ενδεχομένως να συμπεριλάβουμε μέσω τροπολογιών, ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για συστάσεις. Δηλαδή, όταν αναφερόμαστε στη δυνατότητα να προβλέπετε πρόσβαση σε νομικές, δικαστικές αποφάσεις, σε κάποιες αποζημιώσεις για παράδειγμα. Ξέρετε ότι ε, αυτό μπορεί να προβλέπεται σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά πάλι όχι, δεν μπορεί να καταστεί πάντως υποχρεωτικό μέσω της έκθεσης αυτής. Αυτό εναπόκειται, είναι αρμοδιότητα της εθνικής νομοθεσίας. Όσον αφορά ένα ζήτημα το οποίο έθιξαν ορισμένοι συνάδελφοι και που αν δεν κάνω λάθος έχει να κάνει με το σημείο εκείνο που αναφέρεται στα μέλη οικογενειών ελοάδμα. Η έκκληση που κάνουμε εδώ πέρα προς τα κράτη-μέλη ουσιαστικά είναι μια έκκληση που έχει γίνει από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ουσιαστικά δεν λέμε εδώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αλλάξουν το σύνταγμά του για το πώς προσεγγίσουν μια οικογένεια. Προφανώς δεν θα ζητούσαμε ποτέ κάτι τόσο φιλόδοξο. Αλλά όσον αφορά τα μέλη οικογένειας και το συγκεκριμένο αυτό ορισμό, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα προκύπτουν κάποιες συνέπειες. Όταν ένα μέλος της οικογένειας αυτής υποστεί ένα ατύχημα εργασιακό ή ασθενήσει και χρειαστεί τη βοήθεια και την υποστήριξη άλλου μέλους της οικογένειας, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε προκειμένου ποιος αποτελεί μέλος της οικογένειας και ποιος όχι. Όσον αφορά τέλος τα δεδομένα, τη συλλογή των δεδομένων και ολοκληρώνω με την παρατήρηση αυτή, ξέρετε ότι υπάρχουν υπηρεσίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συλλογή των δεδομένων. Καλούμε λοιπόν να συλλέγουν και αυτές δεδομένα και πρόκειται να το πράξουν, αλλά λέμε επίση ότι είναι πολύ σημαντικό και σε εθνικό επίπεδο να γίνεται μια αντίστοιχη συλλογή δεδομένων. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε τελικά να δούμε ποια πρόοδο τελικά σημειώνεται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την καταπολέμηση των διακρίσεων. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε τελικά να προωθήσουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα ευαισθητοποίηση. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ και προσβλέπω σε περαιτέρω συνεργασία με του συναδέλφου. Σας ευχαριστώ όλους. Προθεσμία για την καταβολή τροπολογιών είναι η 3η Μαρτίου το μεσημέρι. Εξέταση των τροπολογιών 22 με 23 Μαρτίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης θα πραγματοποιηθεί 18-19 Απριλίου. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 11 της ημερησίας διάταξης, ε, τη στρατηγική για την ενιαία αγορά. Πρόκειται για πρώτη εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, για την ε, έκθεση πρωτοβουλίας της ΙΜΚΟ για τη στρατηγική για την ενιαία αγορά και θα δώσω το λόγο στην και Τρεμπέσιους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εσωτερική αγορά ε, εάν εφαρμοστεί σωστά, θα δώσει τεράστιες ευκαιρίες ε, στις επιχειρήσεις ε, τα, για τα αγαθά για τα κεφάλαια και έτσι θα δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. Προσπάθησα με τη γνωμοδότηση αυτή να επικεντρωθώ σε κάποια ε, σημαντικά σημεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα για την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, τον τελευταίο καιρό έχουμε κάνει πολλή δουλειά πάνω στον τομέα αυτό, για παράδειγμα με τη γνωμοδότησή μας για την ψηφιακή εσωτερική αγορά. Ως συντάκτη της παρούσας νομοδότησης προσπάθησα να βασιστώ σε αυτά που ήδη έχουμε κάνει εδώ πέρα. Έψαξα να βρω που μπορεί να επιφέρει προστιθέμενη αξία η ευρωπαϊκή αγορά ε, όσον αφορά την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δυστυχώς ήταν ε, περιορισμένος αριθμός λέξεων που μπορούσα να χρησιμοποιήσω, έτσι δεν είχα πάρα πολύ χώρο. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να αναφερθώ στα επιμέρους θέματα. Στις παραγράφους 1, 2 και 3 προσπάθησα καταρχάς να περιγράψω την εξέλιξη της ενιαίας αγοράς. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ενιαία αγορά έχει φέρει ευκαιρίες, ε, υπάρχουν όμως ε, πτυχές που θα πρέπει να βελτιωθούν για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα μέγιστα ε, την ενιαία αγορά για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Στις παραγράφους 3, 4 και 6 αναφέρω ότι είναι σημαντικό να, να γίνει εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για την ε, προστασία κατά, τον, ε, κατά της κατάχρησης των προτύπων. Ε, στην παράγραφο 5 αναφέρω την σημασία δημιουργίας του κατάλληλου πλαισίου. Θέλουμε να προωθήσουμε ένα περιβάλλον όπου να μπορούν να μεγαλώσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να είναι και η δυνατή δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι υπάρχοντες μηχανισμοί θα πρέπει να βελτιωθούν ώστε να προωθείται και εδώ η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Στις παραγράφους 7 και 8 και 9 προσπάθησα να δω την προοπτική την κοινωνική της ενιαίας αγοράς και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει η κοινωνική αντιμετώπιση της ε, αγοράς ε, των υπηρεσιών. Δεύτερον, αναφέρω μέτρα σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες πλαισίου για παράδειγμα όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Τέλος, ε, καλώ την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να, στηρίξουν ε, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, θεσπίζοντας ε, και κατάλληλες διασφαλίσεις για να προστατευτούν τα υπάρχοντα πρότυπα επειδή όπως σας είπα ε, ήταν, υπήρχε περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των λέξεων, δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω τίποτα άλλο στο περιεχόμενο. Ελπίζω όμως ε, με την ε, ενσωμάτωση τροπολογιών των σκιωδών εισηγητών να μπορούμε να διατυπώσουμε μία σαφή θέση. Προσλέπω στις ανταλλαγές που θα έχω με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ σκιώδης απουσιάζει. Δεν ξέρω. Ποιος τον εκπροσωπεί κανείς. Καλά. Να πάμε στη Μαρία Ρενά τότε, σκιώδη ηγήτρια από σοσιαλιστές και δημοκράτες. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Συγήτρια για την έκθεσή σας αυτή, η οποία ευτυχώς έρχεται να εισαγάγει την έννοια του εργαζομένου στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ε, Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Γιατί σχεδόν είχαμε ξεχάσει ω την εσωτερική αγορά, είχαμε και κάτι εργαζομένους εκεί πέρα. Ε, και έχει σημασία η δική μα Επιτροπή να γνωμοδοτήσει και να ασχοληθεί με τους εργαζομένου. Δηλαδή από αυτή τη σκοπιά να το βλέπουμε εμεί στη γνωμοδότησή μα ω Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ για τα διάφορα που προτείνετε. Θα κάνουμε και κάποιε τροπολογίε για να τα συμπληρώσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι σε μια γνωμοδότηση, σε μια έκθεση είναι περιορισμένο ο αριθμό των χαρακτήρων που μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει. Άρα και το μήκο του κειμένου. Στι αιτιολογικές σκέψει ε, θα θεωρούσαμε σκόπιμο για να μην έχουμε παρεξήγηση ότι τι φταίει στην Ευρώπη γιατί υπάρχει κρίση. Δεν είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι και θυμίζουμε την κρίση του 2008 γιατί τίνουμε να τη λησμονούμε. Αυτή η κρίση μας έχει φέρει εδώ που βρισκόμαστε σε τόσο δεινή θέση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να θυμίσουμε λοιπόν ε, τις επιπτώσεις της κρίσης ε, στην αγορά εργασίας και όχι ότι φταίει η αγορά που δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως δεν λέω ότι δεν χρειάζεται βάθυνση εκεί. Επίσης θα πρέπει να δούμε και να θυμίσουμε ε, την ανεργία που είναι πάρα πολύ υψηλή σήμερα στην Ευρώπη, ε, να μιλήσουμε και για τη φτώχεια. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει με τον εσωτερική αγορά, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και ποιοτικέ, αλλά και με σωστή αμοιβή για να μην έχουμε εργαζομένους φτωχούς. Και θα επανέλθω στις προτάσεις ε, στη συνέχεια για τη σωστή αμοιβή για μια εργασία. Επίσης με τη σύγκληση, την κοινωνική σύγκληση μόνο θα προχωρήσουμε σε περισσότερη και καλύτερη εσωτερική αγορά. Σήμερα έχουμε αποκλήσεις και στην εργασία και στα κοινωνικά και στα περιβαλλοντικά. Χωρίς να μιλήσω για τα φορολογικά που μπορεί να απέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους και να ε, επιτείνουν τις δυσκολίες. Όλα αυτά πρέπει να τα θυμίσουμε. Στις προτάσεις που κάνουμε ε, θα υποβάλουμε, είπαμε, τροπολογίες για να πούμε ότι εμείς είμαστε υπέρ μιας βιώσιμης οικονομίας με ποιοτικέ θέσεις εργασίας όμως. Και όταν γίνεται λόγος για διοικητική απλούστευση, απλοποίηση ή το ρέφιτ στο λεγόμενο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η κοινωνική προστασία ή η προστασία της υγείας είναι εμπόδια στην εργασία θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των κανόνων προς τα πάνω και όχι να κάνουμε εκπτώσεις εκεί πέρα γιατί τα θεωρούμε φραγμούς και εμπόδια στην ενιαία αγορά αυτά τα ζητήματα της προστασίας των εργαζομένων. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό, η αγορά εργασίας θα πρέπει και η ιστορική αγορά να οργανώνεται έτσι ώστε να αποκρούει και να ε, καταπολεμά τον αθέμητο ανταγωνισμό. Να υπάρχει και μια δίκαιη ανάπτυξη χωρίς εκπτώσεις, επαναλαμβάνω και με σεβασμό στους εργαζομένους. Θα κάνουμε λοιπόν αυτές τις τροπολογίες, θα τις υποβάλουμε και βεβαίως πάντα με ένα πνεύμα επικοδομητικό. Ε, Madam Harkin, please. το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος της συναδέλφη, η οποία δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ μαζί μας, η κυρία Λόπες να ευχαριστήσω καταρχά τη συντάκτηρα τη γνωμοδότησης. Στη συνέχεια συνάδελφο, λέει τα ακόλουθα. Συμφωνώ με τα όσα λέει η συγγήτρια και με πολλά από τα σημεία τα οποία θίγει στη γνωμοδότηση αυτή. Συμφωνώ απόλυτα ότι οι φραγμοί επιχειρηματικότητας διασυνοριακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν φραγμού στην απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασία. Όντω συμφωνώ ότι η ψηφιακή αγορά προσφέρει νέε ευκαιρίε και νέε προκλήσει που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τελικά η Ευρώπη θα ανταποκριθεί στις νέες δυνατότητες της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Και συμφωνώ ότι η στρατηγική για την έννοια αγορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαίρομαι επίση που η συντάκτρια τη γνωμοδότηση δίνει μια προτεραιότητα στην ενιαία αγορά υπηρεσιών και ότι θα πρέπει και εκεί πέρα να, κα, να καταβληθούν προσπάθειε για να μην έχουμε φραγμού και εμπόδια. Ο τομέα των υπηρεσιών περιέχει πάρα πολλέ ευκαιρίε, όχι μόνο για να αυξηθεί η επιλογή των καταναλωτών, αλλά και να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση με μειωμένο κόστο για του καταναλωτέ. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο τι θα μπορούσε να γίνει στην πράξη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο θετικό περιβάλλον για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε αυξήσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Καλύτερες λοιπόν ευκαιρίες χρηματοδότησης και ένα πιο ελαφρύ διοικητικό περιβάλλον σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πράγματα τα οποία τα ζητάνε ήδη μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ως προς αυτά λοιπόν θα ήθελα να υποβάλω και κάποιες τροπολογίες. Χαίρομαι πάρα πολύ που η συγκήτρια αναφέρεται στις ψηφιακές δεξιότητες ως πρόκληση στην ψηφιακή οικονομία. Θα ήθελα πραγματικά να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτέ τι ψηφιακέ δεξιότητε και σχετικά με αυτό θα υποβάλω κάποιε τροπολογίε. Εν γέννη θεωρώ ότι το σχέδιο γνωμοδότηση είναι πολύ καλό και αποτελεί πολύ θετική βάση για περαιτέρω συζητήσει. Προσβλέπω λοιπόν στην ερωτική μα συνεργασία για την γνωμοδότηση αυτή. Thank you. Uh, I... Ευχαριστώ. Δεν βλέπω την Παλώμα Λόπε. Um, Από την ΚΟΕ. Δεν ξέρω, άλλο κανεί την εκπροσωπεί. Άρα πάμε στους πρασίνους. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Σε αντίθεση με άλλους, Μάλλον όπως και οι άλλοι εκτιμώ και εγώ την ε, δυσκολία ε, του να συμπυκνώσουμε όλα όσα θέλουμε να πούμε σε νέα σύντομες παραγράφους, αλλά κάποια θέματα που θα θέλαμε να συμπεριληφθούν είναι τα εξής. Όσον αφορά τη συμμετοχική οικονομία, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω ως Επιτροπή. Υπάρχουν ευκαιρίες, θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να υπάρχει και επαρκής κοινωνική προστασία και θα πρέπει να εξετάσουμε και την πτυχή της φορολογίας. Κάποιοι μίλησαν για το θέμα της ποιότητας και κλείνει το μικρόφωνο. Και επίσης όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών, δεν μιλάμε εδώ για τον δημόσιο τομέα, θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές το γιατί πράγμα μιλάμε. Επίσης, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υποβάλει κατευθυντήρες γραμμές ε, όσον αφορά τη συμμετοχική οικονομία. Θα θέλαμε λοιπόν να το εξερευνήσουμε αυτό επίσης. Εξετάζει την ε, δυνατότητα να υπάρξει κείμενο για τον τομέα των οικοδομών, το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Επίσης, ζητώ συγγνώμη, δεν βγάζω τα γράμματά μου, λέει ο Μιλήτρια. Σημαντικό είναι να δούμε πώς ταιριάζουν εδώ τα κοινωνικά και φορολογικά συστήματα με όλα αυτά. Να βεβαιωθούμε δηλαδή ότι όλα ακολουθούν ε, την ε, δυνατή διεύρυνση που μπορεί να υπάρξει εδώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ατζέα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την συνάδελφο, την εισηγήτρια, για αυτό το πρώτο σχέδιο γνωμοδότησης το οποίο μας υπέβαλε, ένα πρώτο έγγραφο εργασία ουσιαστικά, το οποίο βέβαια θα τροποποιηθεί με τις δικές μας εστροπολογίες με την ε, γενικότερη επιθυμία να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερα σημεία σε μια γνωμοδότηση η οποία πρέπει να μείνει ευσύνοπτη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνουμε να ελοποιήσουμε κάτι το οποίο θα έπρεπε ουσιαστικά να έχει προγραμματιστεί και να έχει υλοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ με την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς, η οποία ακόμα δεν είναι ενία. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, μετά όσα τα οποία προβλέπουμε, δεν θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε όλες αυτές τις εξωτερικές πιέσεις, οι οποίες θα φτάνουν όλο και πιο δρυμύτερες από τις αναδυόμενες οικονομίες και οι οποίες θα πλήξουν όλο και περισσότερο στο μέλλον την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία θα έχουμε αυτή την ενιαία αγορά. Μια ενιαία αγορά η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή κοινέ ρίζε, δεν έχει κοινό φορολογικό σύστημα, δεν έχει κοινέ εργασιακέ προποθέσει. Δεν είναι ισότιμη για όλους τους εργαζομένους. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όσο θα θέλαμε με την ενιαία αυτή αγορά ή όσο θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει αν πραγματικά εξ αρχής είχαμε προβλέψει διαφορετικές προϋποθέσεις και μια πιο ισχυρή βάση που να μπορεί να μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές πιέσεις. Το ντάμπινγκ, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταφέρνουμε να το αποφύγουμε ούτε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα γίνει όταν θα φτάσουν οι κινέζικες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θα αρχίσουν να χτυπάνε την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα επηρεάσουν το επιχειρησιακό ιστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, όσον αφορά την μετακατάσταση των επιχειρήσεων, ούτε και αυτή καταφέραμε να την αποφύγουμε, γιατί δεν είχαμε δημιουργήσει πάλι την απαραίτητη βάση που θα προέβλεπε τη διατήρηση της βιομηχανικής παραγωγής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έγινε η απαραίτητη δουλειά δηλαδή σε εσωτερικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάναμε απλώς μια επιφανειακή εργασία. Εγώ Πιστεύω ότι η αρχική πρόθεση ήταν θετική, είναι αναγκαιότητα νέα αγορά, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν δημιουργήσαμε γερά θεμέλια. Δεν έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή βάση. Πάρα πολλά πράγματα κανονικά θα έπρεπε να εξετάσουμε. Υφίστανται πολλές διαφορετικές πτυχές αυτή τη στιγμή στην ενιαία αγορά. Πάρα πολλές επικρίσεις θα μπορούσαμε να κάνουμε σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Αν όμως είχαμε ξεκινήσει με μια πολύ πιο γερή βάση, με πολύ πιο γερά θεμέλια, τότε θα είχαμε και μια πολύ πιο ουσιαστική ενιαία αγορά. Θα είχαμε κοινού τότε κανόνες, κοινέ προποθέσει οικονομική ανάπτυξη, και ενδεχομένω ακόμα και ένα ενιαίο νόμισμα το οποίο δεν θα είναι μόνο νόμισμα με οικονομική νομισματική πτυχή, αλλά θα, είναι ένα, θα ήταν ένα νόμισμα το οποίο θα λειτουργούσε πολύ πιο δίκαια για όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Αν είχαμε τη γερή αυτή βάση θα είχαμε και απασχόληση, θα είχαμε αντιμετωπίσει το dumping, θα έπρεπε να είχαμε κανονικά και κοινού φορολογικού κανόνε και κατά αυτόν τον τρόπο θα είχαμε δημιουργήσει μια αγορά εργασίας επιτυχή και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, μια αγορά εργασίας η οποία τελικά οδεύει προς την αποτυχία. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πάρα πολλά προβλήματα που εκκρεμούν ακόμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ντομινίκ Μαρτά εκπροσωπεί την κυρία Μπιζότο. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Να σας πω τι λέει η κυρία Πιτσότο εδώ και ζητεί συγγνώμη για την αποσία της. Για αυτή τη στρατηγική για την ενιαία αγορά και σας διαβάζω. Το 2000 η στρατηγική της Λισαβόνας πανηγυρικά ανακοίνωνε ότι μέχρι το 2010 η ευρωπαϊκή αγορά θα ήταν η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναμική παγκοσμίω. Βρισκόμαστε στο 2016 και οι νέοι μας αλλά και οι γονείς τους είναι άνεργοι, οι πατεράδες τους. Κλείνουν οι επιχειρήσεις γιατί στενάζουν υπό το βάρος του του ανταγωνισμού τη φορολογία, την έλλειψη ελκυστικότητας λόγω ενός κακού νομίσματος του ευρώ. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η στήρα προπαγάνδα και αυτές οι στρατηγικές να τερματιστούν. Τα κράτη θα πρέπει να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές και να φροντίζουν τη βιομηχανία τους, τους ε, ε τεχνίτες τους ε, και τους εργαζομένους, τους εργάτες. Θα έλεγα προσωπικά ότι συμφωνώ και εγώ. Μια ενιαία αγορά μπορεί να πεζότανε ε, με 8. Αλλά επειδή ε, εδώ θέλουμε, ε, ενώ είμαστε βάτραχοι, να είμαστε πιο χοντροί από βόδια, δηλαδή από 8 γίναμε 28, ε, δεν γίνεται να έχεις ενιαίο νόμισμα με 28 χώρες. Ευχαριστώ. And the last word. Ευχαριστώ και το τελευταίο λόγο από πλευράς Κοινοβουλίου. Α, όχι, πρώτα ο κύριος Σούλτσε και μετά εσείς, παρακαλώ. εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μαρτά που ανέφερε το ευρώ γιατί παραλίγο να νομίζω ότι μιλούσε για τη Βόρεια Κορέα. Γιατί τουλάχιστον Ευρώπη εγώ δεν αναγνώρισα στα λεγόμενά του. Εγώ που δεν είμαι σκιώδης ε, για το ΕΛΚ θέλω να μιλήσω για ένα σημαντικό θέμα, αν μου επιτρέπετε, και αυτή είναι η ε, συμμετοχική οικονομία, shared economy. Έγραψε μερικά λόγια και η συγγήτρια. Προφανώς δεν μπορεί να επεκταθεί γιατί έχει περιορισμού στο μήκος της ε, γνωμοδότησης. Τις επόμενες εβδομάδες θα επεκταθούμε αυτή η οικονομία έχει πολλά πλεονεκτήματα σε περίπτωση αμφιβολιών και μπορεί να δημιουργήσει και πολλές θέσεις εργασίας και να αναπτύξει περισσότερο την οικονομία μας το στο Uber ή Airbnb, οι άνθρωποι ίδιοι γίνονται επιχειρηματίες και θα πρέπει να προσέξουμε γιατί οι νόμοι μας δεν είναι ακόμα προσαρμοσμένοι και πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Αυτό ισχύει για την προστασία της εργασίας αλλά και για τη φορολογική νομοθεσία. Θα πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ως στόχο να προωθήσουμε τη βιομηχανική παραγωγή και να δώσουμε περισσότερο χώρο στη βιομηχανία και στην παραγωγή μας στην εθνική οικονομία της κάθε χώρας. Ενώ εδώ την επαναβιομηχάνηση, δηλαδή ε, προϊόντα περίπλοκα τεχνικά που ξέρουμε πολύ καλά στην Ευρώπη να φτιάχνουμε. Και ε, ε, εκεί είναι μια ολόκληρη αλυσίδα παραγωγής αξίας με προμηθευτές, με πάρα πολλές μικρές εταιρείες και χρειάζονται και καταναλωτές αυτοί για να πουλάνε τα προϊόντα τους και εκείνοι να τα αγοράζουν. Και ε, αυτή λοιπόν η αλυσίδα παραγωγής αξίας θα πρέπει να διατηρηθεί γιατί η παραγωγή ενός προϊόντος είναι πάντα πολύ πιο περίπλοκη και δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας από την παροχή υπηρεσιών. Αυτό φέρεται και με τη συμμετοχική οικονομία και πόσο δύσκολο είναι με τέτοια επιχειρηματικά μοντέλα να βγάζουν λεφτά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλέ εταιρείε που είχαν καλέ ιδέε αλλά δεν μπόρεσαν να τι εφαρμόσουν στην πράξη. Αυτή λοιπόν η συμμετοχική οικονομία θα είναι ένα λιθαράκι για να χτιστεί ο τείχο τη οικονομία των υπηρεσιών ε, αλλά θα πρέπει να την ε, πλαισιώσουμε με νόμου και με ε, ρυθμίσει για να ενταχθεί στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Η κυρία Τρεμπέσιος έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γεώδεις συγητές θερμότατα για την τοποθέτησή τους και την τόσο εκτενή στην παρθενική μου έκθεση. Βεβαίως καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε και τα δύο στοιχεία, να μην σκεφτόμαστε μόνο τους εργοδότες αλλά και τους εργαζομένους αλίμονο. Συμφωνώ απολύτως και σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ για τις προτάσεις σα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην έχουμε υπερβολικές ρυθμίσει και υπερβολικές επεμβάσει. Και εντάξει θα πρέπει να σκεφτόμαστε και ε, την αρχή της επικουρικότητας όταν μιλούμε για κοινή φορολόγηση. Παρόλα αυτά τα όσα ωραία λέμε εδώ πέρα, ε, να μην το παρακάνουμε και να μην καούν και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για τις τροπολογίες που θα μου υποβάλλετε. Θα τις δω και από κοινού θα έχουμε χρόνο να εκπονήσουμε μια καλή έκθεση και ισορροπημένη. Σας ευχαριστώ όλους σας για τη συνεισφορά σας. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας και για τις παρουσιάσεις σας. Προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι... 23 του μηνός, Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, μέρα Τρίτη. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 22 με 23 Μαρτίου, ενώ στην Επιτροπή μκο που είναι αρμόδια επί της ουσίας, Απριλίου παρακαλώ. We move on to the next... Και πάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι το 12 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας του Συμβουλίου 2010 Κουλουπού Κουλουπού της 8 Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας πλησίου για τη γονική άδεια και ακολουθούν οι οργανώσεις. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μαρία Αγρινά για να μας πει για ποιο λόγο μας απασχολεί αυτό το θέμα και με ποιον συνεργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, η οδηγία για τη γονική άνθεια είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα οδηγία, γιατί προκύπτει ουσιαστικά από εργασία που κάνανε οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι θέλουν να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές διακρίσεων κατά των γυναικών στο χώρο της εργασίας και ξέρετε ότι το είπαμε οι γυναίκες είναι πολύ συχνά θύματα διακρίσεων, πολλαπλών διακρίσεων στο χώρο απασχόλησης. Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι θέλανε καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και μια καλύτερη κατανομή των καθηκόντων ανάμεσα σε μητέρες, πατέρες, στα πλαίσια του ζευγαριού δηλαδή, όσον αφορά τα οικιακά και όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών. Η Eurofound προχώρησε σε μία μελέτη, μία ανάλυση, σύμφωνα με την οποία η οδηγία αυτή αποτελεί τελικά αποτυχία εν μέρη, διότι όσον αφορά την κατανομή αυτή των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους γονείς ένα 2,7% μόνο των πατέρων χρησιμοποιούν τη δυνατότητα αγωνικής άδειας, επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει τον αρχικό μας στόχο σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, τέτοιες τεράστιες αποκλήσεις. όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρησιμοποίησης της γονικής άδειας από τους πατέρες. Η Eurofound συνδέει το επίπεδο αποζημίωσης της γονικής άδειας με το, δικαίω, με το ποσοστό χρησιμοποίησης της άδειας αυτής από τους πατέρες. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κάνουμε εδώ πέρα κάποιες τροποποίησεις για την οδηγία αυτή. Η οδηγία για την γονική άδεια βέβαια ασχολείται και με το ζήτημα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εργαστούμε και με την Επιτροπή Γυναικών για αυτό το ζήτημα. Επίσης όσον αφορά πάλι την έκθεση για τη γονική άδεια 201 ήταν τροπολογίες που έλαβα. Η ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών ήταν 14 Ιανουαρίου του 2016. Περισσότερες τροπολογίες ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα της μεταβασιμότητας της γονικής αυτής άδειας. Πάλι αποκλείουν πάρα πολύ τα συστήματα μεταξύ τους. Άρα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με την μεταβασιμότητα, με τον μεταβάσιμο αυτό χαρακτήρα των αδειών, της γονικής άδειας. Ξέρετε ότι στις πιο παραδοσιακές νομοθεσίες βλέπουμε ότι η γυναίκα παραμένει στον παραδοσιακό της ρόλο, ενώ οι πιο προηγουμένες χώρες στην κατανομή των καθηκόντων στο ζευγάρι, για παράδειγμα στις σκανδιναβικές χώρες, βλέπουμε ότι χάρη στη μεταβασιμότητα της γονικής άδειας υπάρχει καλύτερη κατανομή των καθηκόντων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρα πρέπει να βρούμε και εδώ τη σωστή εξισορρόπηση Πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη μεταβασιμότητα να μην περιορίσουμε τη γυναίκα σε ένα συγκεκριμένο ρόλο, αλλά να μην εμποδίσουμε ορισμένε χώρε όπω οι σκανδιναβικέ χώρε να προωθήσουν το εθνικό του μοντέλο, το οποίο πιστεύω ότι είναι θετικό και θα πρέπει να προωθηθεί περισσότερο. Μια δεύτερη ομάδα τροπολογιών έχει να κάνει με το ζήτημα τη ε, αμοιβή που προβλέπεται στη γονική άδεια, όπω το λέει και η Eurofound, είναι πολύ σημαντικό να είναι υψηλή αυτή η αμοιβή τη άδεια. Αυτό πιστεύουν και οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να δούνε πώς αυτή η αμοιβή της γονικής άδεια θα μπορέσει τελικά να δοθεί, σε ποιους, για ποια χρονική περίοδο, σε ποιο επίπεδο κτλ. Πάντως το ζήτημα αυτό φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικό προκειμένου να έχουμε αυτή την κατάλληλη κατανομή των καθηκόντων. Έπειτα η διάρκεια της γονικής άδεια. Η διάρκεια δηλαδή όσον αφορά τους διαθέσιμους μήνες στα πλαίσια της άδεια αυτής, αλλά και η διάρκεια όσον αφορά την ε, ηλικία των παιδιών. Δηλαδή, αυτή η γονική άδεια θα πρέπει να ολοκληρώνεται το παιδί φτάνει τα 8 έτη. Δεν θα πρέπει ενδεχομένω να θεωρούμε ότι ένα παιδί χρειάζεται την υποστήριξη των γονιών του και κατά τη διάρκεια τη εφηβεία. ή ακόμα πολύ περισσότερο τότε ότι θα πρέπει να υπάρχει παρουσία των γονών και επομένω γονική άδεια. Επομένω, μα ενδιαφέρει και η περίοδο διάρκεια τη ε, γονική άδεια, αλλά και η σχετική ηλικία του παιδιού. Κάποιες άλλες τροπολογίες σχετίζονται με την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματική ζωής. Και ένα άλλο ζήτημα είναι αυτή η ρήτρα αναθεώρηση τη οδηγία. Έχουμε και γι' αυτό κάποιε τροπολογίε. Όπω σα είπα, 201 συνολικά τροπολογίες τροπολογίε που κατατέθησαν. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να καταλήξουμε σε 21 συμβαστικές τροπολογίες και να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι αφενός υπέβαλαν τις τροπολογίες αυτές και από την άλλη τώρα συνεργάζονται προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε στις συμβαστικές αυτές λύσεις. Προβλέπονται τρεις συνεδριάσεις, 25 Φεβρουαρίου, 1 Μαρτίου και 8 Μαρτίου και πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Για μια φορά σε ευχαριστώ πολύ για την εργασία που έχει γίνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε συνεχίσουμε την εργασία προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο θα εκπροσωπεί όλες τις διαφορετικές απόψεις για έναν κοινό στόχο, καταπολέμηση των διακρίσεων και καλύτερη κατανομή των καθηκόντων ανάμεσα στους δύο γονείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χέκμαν, πρώτος και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, κοιτάω τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην ε, έκθεση αυτή και βλέπω ότι ορισμένες ξεχωρίζουν. Υπάρχουν κάποια θέματα που επαναλαμβάνονται και έρχονται ξανά και ξανά. Δηλαδή και τα θέματα που ανέφερε μόλις η συζήτρια απασχολούν πολλές από τις τροπολογίες για τη μεταβιβασιμότητα ας πούμε, της γονικής άδειας. Εγώ θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Κατανοώ απολύτως τις προθέσεις των συναδέλφων που κάνουν τις τροπολογίες αυτές και τονίζουν την έλλειψη ευκαιριών για τη μεταβιβασιμότητα. Εντάξει, αλλά επαναλαμβάνω το κατανοώ, αλλά φοβούμε ότι μια τέτοια πρόταση θα μπορούσε να έχει αρνητικέ συνέπειε, ε, ιδιαίτερα για εκείνου που θέλουμε να βοηθήσουμε και που μα νοιάζουν περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε τι επιδιώκουμε, τι θέλουμε να επιτύχουμε με τις τροπολογίες αυτές. Θέλουμε να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη περίοδος της γονικής άδειας ή να έχουμε ένα μηχανισμό που να φέρνει ε, την ισορροπία στην οικογένεια και να είμαστε βέβαιοι ότι οι γονείς ε, μπορούν εξίσου να ασχολούνται με το παιδί τους, να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, η υπόθεση αυτή, αν μπορεί να μεταβιβάζεται η γονική άδεια, τότε πολλοί περισσότεροι πατέρες θα θέλανε να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία και να πάρουν εκείνη άδεια. Όχι μητρική δηλαδή, αλλά γονική άδεια από τον πατέρα. Σε πολλές περιπτώσεις η γονική άδεια θα μπορούσε ενδεχομένω να αποβεί και εις βάρος του παιδιού, αν γίνει με λάθος τρόπο. Βεβαίως θα πρέπει να ε, γίνει πολλή δουλειά για να ε, διαφημιστεί η γονική άδεια ε, προς τους πατέρες και όχι να, να τους υποχρεώνουμε να παίρνουν γονική άδεια χωρίς να το θέλουν, γιατί μπορεί έτσι αυτό να είναι εις βάρος του παιδιού, του νεωτέρου μέλους της οικογένειας. Χρειάζεται ένας μηχανισμός πολύ πιο περίπλοκος και να αποφασίζει ο πατέρας αν θέλετε. Ε, και είναι κατά περίπτωση ε, ποιος θα παίρνει την άδεια. Λοιπόν, εξετάζεται αν θα είναι μόνο η μητέρα και οι δύο γονείς. Δυστυχώς δεν μπορώ εγώ να συμφωνήσω με την ιδέα που λέει ότι θα πληρώνεται και θα μείβεται 100% αυτή η άδεια. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί για να μην πω ανεφάρμοστο. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Κοιτάξτε τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Στην αναθεώρηση της οδηγίας για τη μητρική άδεια είδαμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήταν τεράστιο πρόβλημα για σφιχτούς προπολογισμού σε τέτοιους καιρούς. Πολύ καλύτερο θα ήταν να έχουμε μια λύση πιο ευέλικτη. Παράδειγμα, να σας δώσω το παράδειγμα της Πολωνίας. Έχουμε μητρική άδεια ε, αμοιβόμενη εξάμηνη στην Πολωνία. Και μετά από αυτό υπάρχουν έξι μήνες ε, γονικής άδειας όπου ένας από τους δύο γονείς παίρνει το 60% της αμοιβή του και μπορεί να το μεταβιβάσει ε, και να το μετατρέψει σε αμοιβόμενη κατά 80% πλέον άδεια. Αυτή η λύση νομίζω είναι καλή και θα μπορούσε να αποτελέσει και παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής. Πολλές από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί έχουν να κάνουν και με τα προβλήματα της ορολογίας. Και εδώ πραγματικά έχουμε να διαδραματίσουμε ένα ρόλο για να εναρμονίσουμε την ε, ορολογία που χρησιμοποιούμε και να γίνει αυτή συστηματική. Γιατί δεν κάνουν όλες οι χώρες διάκριση ανάμεσα στη μητρική, πατρική και γονική άδεια. Και αυτό μας δυσκολεύει έτσι περαιτέρω τη ζωή μας. Επίσης, να σκεφτούμε και το θέμα της επιστροφής στην εργασία μετά από τη μακροχρόνια απουσία λόγω άδειας. Όταν επιστρέφουν στην αγορά εργασίας οι γονείς, χρειάζονται και οι δύο γονείς και το ίδιο το παιδί ιδιαίτερη προσοχή. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα λέτε. Από τη σκοπιά μου λοιπόν, το σημαντικότερο ζήτημα εδώ της έκθεσης ή τα σημαντικότερα ζητήματα καλύπτονται. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι θα συνεργαστούμε καλά με την εισηγήτρια και με τους γεώδεις συγητές και θα βρούμε συμβιβαστικές λύσεις που θα ικανοποιούν τους πάντες. Και το αποτέλεσμα θα είναι καλό και λογικό. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Gericke, e Ευχαριστώ, κύριο Γκέρικε, σκιώδη ηγητής από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Αρένα για την έκθεση της ε, σχετικά με την γονική άδεια και θα ήθελα να επαναλάβω ότι ε, το διάστημα που μεγαλώνει κανείς τα παιδιά του δεν είναι άδεια. Εγώ επί χρόνια συμμετείχα στην ανατροφή των παιδιών μου. Πρόκειται για δουλειά. Ε, σκεφτείτε ότι στα νηπιαγωγεία θεωρείται εργασία. Δεν είναι λοιπόν διακοπές. Όποιο θεωρεί λοιπόν ότι ο χρόνο ανατροφή είναι άδεια, μήπως μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή, λέει η πρόεδρο έχουμε πρόβλημα με τη διαρμηνία. Σας παρακαλώ, ξεκινήστε από την αρχή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ την συνάδελφο Αρένα για την έκθεσή της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 Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα λειτουργεί. Μπορεί να είναι τεχνικό πρόβλημα, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. <clears throat> Ο τεχνικός το εξετάζει. Δώστε του δύο λεπτά. Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα με γαλλική διερμηνία τον κύριο Γκέρικε. Τέταρτη φορά θα ξεκινήσω, λέει ο, ο μιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ την συνάδελφα Αρενά για την έκθεσή της, ε, για την, για την έκθεσή της και θα ήθελα να τονίσω ότι ο χρόνος ανατροφής των παιδιών δεν είναι άδεια, δεν είναι διακοπές. και εγώ είμαι πατέρας 7 παιδιών και επί 10 χρόνια συμμετείχα στην ανατροφή των παιδιών μου ο χρόνος ανατροφής είναι δουλειά, είναι εργασία. Στα, στους παιδικούς σταθμούς και στα νηχαγωγεία θεωρείται δουλειά. Δεν είναι λοιπόν διακοπές για τους γονείς. Σας παρακαλώ λοιπόν να διαγράψουμε τη λέξη αυτή από το λεξιλόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κανείς δεν μιλάει πια για διακοπές των γονέων. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε Ε, να ε, αλλάξει την κατάσταση διότι και εγώ ήδη από την αρχή της θητείας αυτής είπα ότι χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα στο θέμα αυτό και έχω τρία βασικά αιτήματα. Καταρχάς, ας ε, συνεννοηθούμε, ε, ας έχουμε κοινού όρους, ας δεχτούμε την ποικιλομορφία των συστημάτων, να βρούμε λεξιλόγιο ε, για την προστασία της μητρότητας. Δεύτερον, την οδηγία για την προστασία της μητρότητας, ας την αφήσουμε στα χέρια της Γενικής Διεύθυνσης για την Απασχόληση απασχόληση. διότι η μεταφορά του θέματος αυτού σε άλλη υπηρεσία θα σημαίνει και αποδυνάμωση του θέματος αυτού. Τρίτον, ας εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους ακούσουμε όταν μας παρουσιάσουν τις ιδέες τους ε, για νέα οδηγία για την ε, προστασία της μητρότητας ε, και, και μάλλον είμαι πολύ πρωτοπόρος εδώ, μήπως θα ήταν χρήσιμο η οδηγία να βασίζεται στο άρθρο 152 της συνθήκης. Αυτό μπορεί να σας εκπλήσει από το στόμα ενός Ευρωβουλευτή, αλλά η διαδικασία ε, κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι απλά ένας παρατηρητής στο περιθώριο. Ε, νομίζω όμως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαδικασία αυτή ε, θα ήταν ένα σημαντικό βήμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν από το Άλτε σκιώδη εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ την εισηγήτρια και συμφωνώ απολύτω ε, με την ε, σύνοψή σας ε, σχετικά με τους τέσσερις τομεί, του οποίους θα πρέπει να εξετάσουμε στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Όσον αφορά τι τροπολογίε τη ΑΛΔΕ, έχουμε το θέμα της μεταβασιμότητας σύμφωνα με την οδηγία του 2010 έχουν δικαίωμα οι εργαζόμενοι σε γονική άδεια ε, και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι πατέρες να συμμετέχουν στην γονική άδεια και πιστεύω ότι συμβάλλει αυτό στην ισορροπία ε, εργατικού και ε, ιδιωτικού βίου και για τους άντρες και τις γυναίκες. Ακούω αυτά που είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην ε, χαλάσουμε τα ε, καλά εθνικά συστήματα αλλά θα πρέπει να ε, έχουμε και νομισμό στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Δύο βασικά θέματα θέλει να αντιμετωπίσει αυτή η νομοθεσία. Πρώτον, ε, η ισότητα ε, ανδρών και γυναικών και δίκαιη ε, κατανομή των εργασιών ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες και να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Και βλέπουμε ότι ο στόχος του 75% όπως προβλέπεται στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 για τις γυναίκες ε, εκπληρώθηκε στο, το 2014, αλλά ε, για τις γυναίκες το ποσοστό είναι 63%. Γνωρίζουμε ότι η, ε, ότι οι υπηρεσίες φύλαξης των παιδιών αποτελούν σημαντική προϋπόθεση. Και είναι σημαντικό και το θέμα της αποσμίωσης, διότι δεν μπορούμε από τη μία να λέμε ότι θέλουμε ευελιξία, από την άλλη όμως και να έχουμε αυστηρούς κανόνες για τη μη μεταβασιμότητα, αλλά από την άλλη να μην είναι ελκυστικό για τους πατέρες να πάρουν γονική άδεια. Νομίζω λοιπόν ότι τα επίπεδα αποζημίωσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Ε, σημαντικό ρόλο παίζουν και άλλα θέματα όπως είναι η ευελιξία του συστήματος αδειών, η ευελιξία των ε, υπηρεσιών φύλαξης ε, των παιδιών και βέβαια πολλοί κόσμοι φοβάται και τι θα γίνει όταν επιστρέψει πάλι στην αγορά εργασίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν ε, την απόφαση πατέρων να πάρουν γονική άδεια ή όχι. Νομίζω ότι το θέμα της αμοιβή ε, θα αποτελέσει κίνητρο μπορεί να θεωρηθεί υποκατάσταση του εισοδήματος ή κάποιου ποσοστού του. Ωστόσο υπάρχουν ε, κάποια σημεία με τα οποία έχω πρόβλημα, διότι εισάγεται την ε, ιδέα ότι θα πρέπει να βασίζεται ε, στο μέσο ποσοστό μητρικής άδειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικά αυστηρό, αλλά πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύση. Και ε, τέλος, σε κάτι το οποίο ανέφερε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ. Έχουμε τρία διαφορετικά συστήματα, ε, μητρική άδεια, και γονική, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να ε, υπάρξει συνδυασμός των τριών συστημάτων αυτών, συγχώνευση, για να έχουμε ένα συνεκτικό σύστημα και μάλιστα σε όλα τα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συμφωνήσω με την ε, ιδέα αυτή και προσλέπω στην καλή συνεργασία με την εισηγήτρια στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Uh, thank Ευχαριστώ. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, έχω χάσει το χαρτί μου πάλι. Ε, από την ΚΟΕΣ και όδηση συγγήτρια. Αποουσιάζει, λέει η κυρία γοζάλης Παγιάς. Αποουσιάζει ο σκιώδης συγγητής μας και δεν μου έχει δώσει και τη θέση του να τη διαβάσω. Έχω εργαστεί εγώ, έχω κάνει τροπολογίες. Αλλά για να μιλήσω εγώ εξ ονόματός μου, να περιμένω όταν ήρθε η ώρα των ε, κανονικών βουλευτών και όχι των σκιωδών. Ωραία. Η κυρία Βάνα είναι εδώ από τους Πρασίνους, όχι. Η ευθυντή από την Λαορατζέα που δεν λείπει ποτέ. τι un premio δύο πρέπει να πάρω, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, συμφωνώ με την τοποθέτηση της Μαρία Ρενά. ότι ήδη και στην προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε κάνει, είχαμε πει και το είχε πει τότε και η συγγήτρια, ότι έχει καθυστερήσει σε πολλές χώρες, όπως και στην Ιταλία, η σωστή εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό νομοθετικό αυτή τη στιγμή και ένα κενό εφαρμοστικό. Και νομίζω ότι θα έχουμε τελικά και ένα πολύ μεγάλο χάσμα, δηλαδή διστάμενες απόψεις. Προφανώς η οδηγία αυτή θέτει κάποια ζητήματα τα οποία είναι προβληματικά. Νομίζω λοιπόν ότι για αυτά πρέπει να γίνει μια συζήτηση, δεν υπάρχει σύμπνοια αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς υποβάλαμε τροπολογίες συγκεκριμένες και ουσιαστικές. Είναι πολύ σημαντικό το πεδίο εφαρμογή, για παράδειγμα, να ισχύει τόσο για τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ότι ε, στον ε, δημόσιο τομέα έχουμε πάρα πολλά συστήματα προστασίας του εργαζομένου, από την άλλη στον ιδιωτικό τομέα ο εργαζομένος είναι πάρα πολύ εκτεθειμένος. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα είναι ποιο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει γονική άδεια για μακροχρόνια περίοδο. Γιατί ξέρετε ότι ε, λέμε εδώ πέρα ότι θα μπορούσε η γονική αυτή άδεια να χρησιμοποιηθεί μέχρι το 12ο έτος του παιδιού. Άμα πρέπει να δούμε όμως αυτό στην πράξη πώς θα χρησιμοποιηθεί και πώς, θα, πώς δεν θα λειτουργήσει κατά του ίδιου του εργαζόμενου. Δηλαδή να αποτελέσει αυτό πραγματικά δικαίωμα το οποίο θα είναι αναφέρετο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η γονική άδεια είναι διακοπές. Δεν θα μπορούσε βέβαια να θεωρηθεί ότι είναι και αναρωτική άδεια. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή οδόνα μας στις δύο αυτές προσεγγίσεις, τη χρυσή τομή. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά, ιδίως όσον αφορά τους άντρες, υπάρχει ένας κάποιος δισταγμός να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γονική άδεια, που εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Και αυτό εξαιτία των εργασιακών προποθέσεων που αντιμετωπίζουν και επειδή φοβούνται ότι θα καταφέρουν να επανανταχτούν στην αγορά εργασίας για μας στην Ιταλία τα όσα προτείνεται αυτή τη στιγμή στη γνωμοδότηση αποτελούν πραγματικά επιστημονική φαντασία. Δεν υπάρχει καν η απαραίτητη νοοτροπία στη χώρα μου προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά, να υλοποιηθεί η οδηγία. Γι' αυτό σα έλεγα ότι τουλάχιστον για την Ιταλία βρίσκεται σε εμβρική ακόμα φάση αυτή η οδηγία. Τώρα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γονική αυτή άδεια εκ παραλίλου με άλλα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται για τους αποσπασμένους για παράδειγμα εργαζομένους ή αυτοί που εργάζονται εκτός της χώρας τους. Παράλληλα να προβλέπεται για τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού να έχουμε χρησιμοποιήσει τις άδειες αυτής. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση με πληθυσμό ο οποίος γυράσκει όλο και περισσότερο, με ένα ποσοστό γονιμότητας το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Νομίζω λοιπόν ότι ε, είναι πολύ σημαντικό και δεδομένων των ε, οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και που σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν την ε, αύξηση της γενετικότητας, να μπορούμε τουλάχιστον να χρησιμοποιούμε αυτή την γονική άδεια και βέβαια να δοθούν και τα κατάλληλα κίνητρα για την αύξηση της γενετικότητας. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει επίση και μία έρευνα για να δούμε πραγματικά πώ εφαρμόζεται αυτή η οδηγία στα κράτη-μέλη, όχι απλώ στατιστικά δεδομένα. Μία πραγματική σφαιρική έρευνα για το πώ εφαρμόζεται, πώ υλοποιείται συγκεκριμένα η οδηγία αυτή σε κάθε κράτο μέλο. Γιατί πραγματικά το πανλαμβάνω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο νομοθετικό κοινό το οποίο μα ανησυχεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ζωέλ Μελά, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Περί τίνος συζητούμε τώρα. Γονική άδεια, μετρική, πατρική, όλα αυτά είναι πολύ περίπλοκα. Για ένα πράγμα πρόκειται. Πώς θα υποδεχτεί μια οικογένεια ένα παιδί. Οικογένεια στην οποία δουλεύουν και οι δύο γονείς. Γιατί έχουν την ηλικία να είναι επαγγελματικά ενεργοί. Αλλά από περίεργες ατραπούς φέρνουμε τη γυναίκα υποχρεωμένη να εργάζεται. Ενώ αν δούμε τι γίνεται στη Γαλλία υπάρχει η ανεργία, πέφτουν οι μισθοί και βλέπουμε ότι σήμερα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο γονείς για να φέρουν τα ίδια χρήματα που έφερνε ο ένας πριν από 20 χρόνια. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί ποια είναι ε, η ευθυνή της Ευρώπης γιατί είναι τηλεκατευθυνόμενη αυτή στη φτώχεια και στη φτωχοποίηση της οικονομίας σε κάθε χώρα. Πέρα από αυτά θα πρέπει να δούμε πώς η, μητέρα υποδέχεται το παιδί στη ζωή της. Και η γυναίκα όπως και ο άνδρας έχουν 24 ε, ώρες ε, στο 24ωρο. Δεν υπάρχει θεωρία του γένους εδώ. Και σκεφτείτε πόση ώρα πρέπει κανείς να κοιμάται, να δουλεύει και να είναι καθοδόν από και προς το σπίτι τη δουλειά. Άρα το μόνο που μένει είναι γονική άδεια. Γονική άδεια είναι ο σωστό όρος, πραγματικά. Γιατί και ο πατέρας και η μητέρα μπορούν να συμμετέχουν στην ανατροφή, δεν μπορούμε ε, να επιβάλλουμε ποσοστώσεις. Η ώρα του πατέρα, ο μήνας του πατέρα, ο μήνας της μητέρας, όλα αυτά είναι ιδεολογικέ αγγυλώσει με τη θεωρία του γένους, όπου τα πάντα είναι ίδια, όλα είναι ανταλλάξιμα και συγκρίσιμα θα τα ξαναπούμε όταν αυτοί οι κύριοι αποκτήσουν τεχνητή μήτρα για να δούμε πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Ε, για να δούμε λοιπόν την αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει να διαφυλαχθεί πριν ε, τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία ή τα ευρωπαϊκά διαβήματα. Εντάξει, γιατί όχι, αλλά υπάρχουν διάφορα κοινωνικά συστήματα, αλλά ε, θα πρέπει να δούμε πόσο κοστίζει αυτό, έτσι, ημερησίως ε, όταν χρειάζεσαι μια νταντά για να φροντίζει το παιδί σου και υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη και διαφορετική κατάσταση, επικουρικότητα. Επίση, η ελάχιστη διάρκεια για μα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιβληθεί άνωθεν. Υπάρχουν επαγγέλματα όπου οι γυναίκε λόγω των διπλωμάτων, των πτυχίων, των δεξιοτήτων του μπορούν κάλλιστα να επιστρέψουν γρήγορα στη δουλειά. Και δεν είναι το ίδιο σε όλα τα επαγγέλματα ή κάποιες άλλες γυναίκες που δουλεύουν σε επαγγέλματα υγείας ή έχουν άλλα προβλήματα υγείας οι ίδιες και δεν μπορούν να γυρίσουν στη δουλειά τους. Le monde du travail, le monde... Θα πρέπει να υπάρχουν γέφυρες που να συνδέουν τον κόσμο της εργασίας με τον κόσμο των σπουδών. Ε, όλα αυτά είναι αλληλένδετα και για να γίνουν όλα αυτά δεν βλέπω ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Υπάρχουν χώρες που έχουν προχωρήσει πολύ στην προστασία ε, της μητρότητας και της γονικής άδειας. Ίσως θα έπρεπε αντίθετα η Ευρώπη να ασχοληθεί με το να είναι λιγότερο δεσμευτική ε, προς τις επιχειρήσεις. Γιατί και επιχειρήσεις έχουν ε, παιδικούς σταθμούς και οι μισθοί δεν θα πρέπει να είναι προς τα κάτω συμπιεσμένοι όπως στην απόσπαση εργαζομένων που δεν υπάρχει καμία απολύτως θέση για τις γυναίκες. Πώς μπορείτε να αποσπάσετε μια γυναίκα όταν θέλετε να, ε, να κάνετε οικογένεια, πού να πάει η γυναίκα να σηκωθεί, να φύγει, να αποσπαστεί. Γιατί γυράς η Ευρώπη, μα βλέπετε γιατί. Ανησυχούν οι Ευρωπαίοι, ανησυχούν, θέλετε να κάνουν παιδιά. Εδώ δεν ξέρουν τι τους γίνεται από πλευράς φορολογικής, οικονομικής, απέναντι και στην τρομοκρατία. Εκεί φτάσαμε. Και οι γυναίκες και οι άνδρες τι να κάνουν οι άνθρωποι, παιδιά θα κάνουν. Ε, παρετούνται και βλέπουμε και να μειώνονται οι πολύτεκνες οικογένειες. Η Ευρώπη καλά θα έκανε λοιπόν να κοιτάξει την αυλή της και να ασχοληθεί με τα δικά της, ναι στη γορική άδεια, αλλά εμπλήρη επικουρικότητη. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, uh, Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαλέτρα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η τελική μεταφορά της οδηγίας αυτής για τη γονική άδεια έληξε το 2013. Οι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπής κάνουν αυτή τη στιγμή αναχώρα έναν έλεγχο τη εφαρμογή οδηγία αυτή και έχουν ανταλλαγή απόψεων με πολλά κράτη-μέλη όσον αφορά την εθνική μεταφορά τη οδηγία αυτή και το πόσο συμμορφώνται τα κράτη-μέλη με αυτή την οδηγία. Όταν ολοκληρωθεί ο διάλογο αυτό με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεκινήσει δικασίε επί παραβάση, σε περίπτωση, αν το κρίνει αυτό αναγκαίο βέβαια. Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομομαθών για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών θα προετοιμάσουν μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Έχει προετοιμαστεί μάλλον η έκθεση αυτή και είναι ήδη διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής για τους εργαζομένους γονείς, μια σημαντική πρωτοβουλία για φέτος, Έχουμε εδώ πέρα μία απόσυρση, όπως ξέρετε, της πρότασης 2008 όσον αφορά την γονική άδεια. Ανταυτού είχαμε ήδη από τον Αύγουστο έναν οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιτευχθεί αυτή η συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Νομίζουμε ότι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε εδώ πέρα μια καλύτερη ισορροπία. Με την νέα αυτή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπουμε στα εξαρτώμενα μέλη, στα παιδιά, να προστατεύονται καλύτερα στα πλαίσια του νέου αυτού κοινοτικού πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να προσαρμόστε περισσότερο στι συνθήκε στην αγορά εργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασία όλων των γονιών, καλύτερη κατανομή των καθηκόντων, των οικιακών καθηκόντων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άλλο ένα στόχο μα. Ο δικό χάρτη αναφέρεται επίση στην προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου προβλέπονται εναλλακτικέ προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε το νομοθετικό πολιτικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον δικό αυτό χάρτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε και δύο διαβουλεύσει. Η πρώτη διαβούλευση είχε να κάνει με του κοινωνικού εταίρου και η δεύτερη διαβούλευση είχε να κάνει με του υπόλοιπου ενδιαφερούμενου φορεί. Ευχαριστώ. Thank you. The last word to the rapporteur, Maria Arena. Μαρία Ρέν έχει το λόγο. Να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για τη συμμετοχή τους αυτή, την πολύ ενεργή συμμετοχή τους, προσπαθώντας και αυτοί να πετύχουν την κατάλληλη ισορροπία. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο απότερο στόχος μας. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εργασία που έχει κάνει και που συνεχίζει να κάνει για την εκπόνηση αυτού του δικού χάρτη και το πιο σημαντικό, όπως το είπατε και εσείς, είναι να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε και τα τρία αυτά νομοθετήματα, άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας και γονική άδεια. Να καταφέρουμε να συμπεριλάβουμε και να συνδυάσουμε και τις τρεις αυτές πρωτοβουλίες, οι οποίες αλλοσυμπληρώνονται. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώ η Ιταλίδα συνάδελφο δεν είναι παρούσα. Πολλέ φορέ υπάρχει μια κάποια σύγχυση όταν μιλάμε για άδεια μητρότητα, άδεια πατρότητα και γονική άδεια. Το είπαμε και πριν από λίγο από αυτό. Υπάρχουν διαφορετικέ διαστάσει με βάση τη χώρα στην οποία κατοικούμε. Πρέπει να σα πω ότι όσον αφορά τη γονική άδεια, η οποία μπορεί να φτάσει τα 12 έτη του παιδιού, δεν πρόκειται για γονική άδεια πλήρη, η οποία θα ξεκινήσει από τότε που θα γεννηθεί το παιδί και θα φτάσει μέχρι το 12ο έτος ηλικία του. Αναφερόμαστε προφανώς σε μια γονική άδεια που ο γονιός θα πάρει, οι γονείς θα πάρουν κατά συγκεκριμένα χρονικά σύστημα, κατά συγκεκριμένα χρονικά κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με συγχωρείτε, μέχρι να φτάσει το παιδί το 12ο έτος ηλικία. Στόχος είναι να καταφέρουμε να συνδυάσουμε το δικαίωμα αυτό με τις συνθήκες εργασίας του ενός ή του άλλου γονιού και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τα παιδιά, ιδίω αυτά τα οποία βρίσκονται σε πιο μικρή ηλικία. Α μην προκαλούμε όμω σύγχυση, έπρεπε να κάνω τη διευκρίνηση αυτή. Δεν μιλούσαμε ποτέ για συνεχιζόμενη περίοδο γονική άδεια μέχρι να φτάσει το παιδί το 12ο έτο ηλικία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τι παρατηρήσει πάντω που κάνατε και είμαι σίγουρο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη πρόταση, εφόσον από ό,τι βλέπει περισσότεροι συμφωνούμε σε κάποιου κοινού στόχου. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Τάνια Κονζάλες, θέλετε και εσείς να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια και τις σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα λίγο να σας πω τι λέει η δική μας αντιπροσωπεία για τις πατρικές άδειες και γονικές και μητρικές. Αυτά είναι ατομικά δικαιώματα. που δεν έχει να κάνει με το κάθε ζευγάρι ή με τη συμβίωση. Σε πολλές χώρες οι άδειε δίνονται ε, κατά το δοκούν και κυρίως οι γυναίκες αναλαμβάνουν την άτροφη των παιδιών και παίρνουν τις άδειε αυτές. Αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες ε, ως προς τη συμμετοχή ε, των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και πολύ συχνά ε, φοβούνται οι επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν γυναίκες γιατί σου λέει θα κάνεις παιδί και μετά θα πάρεις μητρική άδεια και δεν θα μου μείνεις εδώ, θα φύγεις. Ε, με άδεια θα πρέπει να σε πληρώνω κτλ. Και αυτό ε, σημαίνει ανισότητα δικαιωμάτων του πατέρα και της μητέρας στην ανατροφή του παιδιού τους. Και τελικά διαιωνίζεται μία διαρθρωτική ανισότητα που υπάρχει και που πρέπει να καταπολεμήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχει κοινή ανατροφή 100% των παιδιών και των ατόμων των εξαρτημένων από τους γονείς αυτούς. Γι' αυτό οι περισσότερες τροπολογίες μας προς τα εκεί στρέφονται. Και ε, η πατρική άδεια να είναι ίδια με τη μητρική 100% αμοιβόμενη, αλλά χωρίς μεταβιβασιμότητα για να παίρνει και ο καθένα την άδειά του και να μην υφίσταται διακρίσεις η γυναίκα στην αγορά εργασίας. Πολλέ από τι τροπολογίε που κάναμε ε, προ τα εκεί πηγαίνουν. Να δείξουν ότι οι πατέρες, οι άνδρες έχουν ευθύνη κι αυτοί. Και αυτό να έχει ε, πλεονεκτήματα για όλη την κοινωνία που είναι διαφυσβήτητα και όχι μόνο για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας και άλλα πλεονεκτήματα και ε, που να είναι προς όφελος όλης της κοινωνίας. Υποστηρίζουμε λοιπόν και την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για να αυξηθεί και ο αριθμός των υπηακών σταθμών και η ποιότητά τους. Είναι πολιτικές, είναι μάλλον υπηρεσίες που πλήττονται από τις πολιτικές λιτότητες και τις περικοπές για να μπορεί ο κόσμος να δουλεύει και να ανατρέφει και τα παιδιά του. Όλα αυτά τα στοιχεία θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να συμπεριληφθούν στην έκθεση και να ληφθούν υπόψη. Και ουσιαστικά περί τίνος πρόκειται όταν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, είναι πολύ ωραία στα χαρτιά, αλλά ε, διαονίζονται πρακτικές του παρελθόντος που πρέπει να σπάσουν και να καταπολεμηθούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ διευκρίνηση σε σχέση με αυτό το οποίο μόλις τώρα είπατε. Δεν ξέρω αν δεν κατάλαβα καλά από τη διερμηνία και ζητώ συγγνώμη από τη διερμηνείς αν πραγματικά το είπατε αυτό το πράγμα. Είπατε ότι πρέπει να υπερασπίσουμε τα ατομικά δικαιώματα, εξατομίκευση δηλαδή των δικαιωμάτων, δικαιώματα οι άντρε, δικαιώματα οι γυναίκες, πατέρες και μητέρες και από την άλλη είπατε τα δικαιώματα αυτά πρέπει να είναι μεταβιβάσιμα. Υπάρχει μια κάποια αμφισημία σε αυτά τα οποία είπατε. Αυτό όντω είπατε, ενδεχομένω να μην κατάλαβα καλά. Άκουσα τη λέξη μεταφορά, μεταβιβασιμότητα, η οποία δεν συνάδει πάρα πολύ με την αρχική σα παρατήρηση. Όχι, ίσα ίσα να μην μεταβιβάζετε. <laughs> ναι, ναι, να μην μεταβιβάζετε. Όχι, ο καθένα να παίρνει την άδειά του. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόληση θα πραγματοποιηθεί 16 ή 17 Μαρτίου. Του τουλεχθέντος θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αύριο θα ξεκινήσουμε στις 9 το πρωί. Έχουμε δημόσια ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας. Και είναι πολύ σημαντική η ακρόαση αυτή. Έχει να κάνει με, το, με την κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας. και είναι βέβαια ιδιαίτερα επικαιρό το θέμα υπό το φως του προσφυγικού. Ελπίζω λοιπόν ότι θα είναι αθρώα η προσέλευση για να ακούσουμε τους προσκεκλημένους και ελπίζω ότι θα συμμετάσχετε και στη συζήτηση. Και αμέσως ε, μετά από αυτήν την ακρόαση έχουμε μία ώρα σεμιναρίου για τις εξελίξεις όσον αφορά τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, υπό την Τρόικα. Ελπίζω λοιπόν ότι θα παρακολουθήσετε και αυτήν τη συζήτηση, διότι έχουμε πολλές συζητήσεις πάνω και στα δύο αυτά θέματα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε νέα στοιχεία και νέες απόψεις. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Ήταν δύσκολη η ψηφοφορία. Χαίρομαι που κάποιοι επιβιώσαμε ώστε να συμμετάσχουμε και στο δεύτερο μέρος της ε, συνεδρίας της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο.